Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε. Την απογευματινή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ώρα ψηφοφορίας. Θα αρχίσουμε με την ψηφοφορία για την θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 ως 2020. Ξέρω, ξέρω. Έχω να σας πω κάτι, αλλά θα σας δώσω το λόγο μετά. Σήμερα ψηφίζουμε για το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής μας. Συνεισηγητές ο κύριος Λάμπερτ Βανίστελρο και η κυρία Κωνσταντσα Κρέλη για την νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι συνεισηγητές μας ψηφίασαν το σχέδιο έκθεσης του το Σεπτέμβριο. Πρότειναν 58 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Μέχρι την ε, καταληκτική ημερομηνία είχαμε 204 πρόσθετες τροπολογίες που υποβλήθηκαν. 264 τροπολογίες σύνολο από αυτές οι 172 προήλθαν από άλλες επιτροπές. Η Συνδεδεμένη Επιτροπή σύμφωνα με τον κανόνα 54 είναι η ΕΚΟΝ. Ε, υπέβαλε 40 τροπολογίες. Κάποιες από αυτές είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη ΕΚΟΝ. Η Επιτροπή προπολογισμού υπέβαλε 14, Επιτροπή Απασχόλησης 86. Και αυτές ε, σύμφωνα με τον κανόνα 53 συν. Η Επιτροπή Αλίας και η Επιτροπή Πολιτισμού γνωμοδότησαν σύμφωνα με τον κανόνα 53 με 29 και 3 τροπολογίες αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων για το θέμα αυτό, όπως αποφασίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 4 Μαΐου 2016, αρκετές τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή μας ε, βρίσκονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Κάποιες ε, λοιπόν δεν είναι ε, δεκτές από την Ρέτζη, δεν θα τις ψηφίσετε σήμερα. Τις έχετε αλλά δεν θα τις ψηφίσετε και όπως βλέπετε τον κατάλογο ψηφοφορίας που ετοίμασε η Γραμματεία, Θα ψηφίσουμε τα άρθρα 5F έως 7.3α και 3β και τις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 4 της ε, πρότασης της Επιτροπής. Και μετά από εκτενέστατες διαπραγματεύσεις ε, των σκιωδών εισηγητών της Επιτροπής μας, αλλά και των ε, σχεδόν των άλλων επιτροπών, προτείναμε 28 συμβιβαστικές τροπολογίες. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως μετά την τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα θα ψηφίσουμε και για την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την σύσταση διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία θα αποτελείται από την πρόεδρο της Ρέτζη, τους εισηγητές, τους σύνης, ε, μάλλον, τους κοιόδης εισηγητές, έναν εισηγητή σύμφωνα με το άρθρο 54 και μετά ε, την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, των ε, εισηγητών των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Απασχόλησης. Αυτά λοιπόν ε, ως ενημέρωση πριν την ψηφοφορία. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Αλλά η κυρία Ρέντκε ζήτησε το λόγο και ε, παρακαλώ τον έχετε. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν ήθελα να σα διακόψω πιο πριν. Ήθελα όμω να αναφερθώ σε κάτι διαδικαστικό ε, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουμε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να αλλάξει η διαδικασία που ακολουθούμε προς το παρόν. Ακολουθούμε τον κανόνα 73 και θα ήθελα να αλλάξει σύμφωνα με τον κανόνα 59. Αυτό σημαίνει ότι η επί Επιτροπή θα ε, την έκθεση στην Ολομέλεια και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας εκθέσω τους λόγους μου γιατί πιστεύω πως αυτή η διαδικασία είναι καλύτερη. Καταρχάς, εάν έχουμε μια ισχυρή εντολή από την Ολομέλεια για την έκθεση αυτή, θα ενισχύσει τη θέση του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο απέναντι στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δεύτερον, όπως αναφέρατε κι εσείς, υπάρχουν αρκετές επιτροπές που εμπλέκονται είτε με γνωμοδοτήσεις είτε με αποκλειστική αρμοδιότητα όπως η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Εάν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε ακόμα καλύτερα τις γνωμοδοτήσεις και τις προτάσεις των άλλων επιτροπών και να έχουμε ευρύτερη στήριξη. Τρίτον, ε, αναφέρθηκε το επιχείρημα ότι χρονοτριβούμε γιατί ακριβώς έχει περάσει πολύς καιρός για το θέμα αυτό, αλλά ε, μια που θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο, έχουμε ακόμα και την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και την Ολομέλεια του Ιανουαρίου για να ψηφίσουμε ε, όλοι. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τη διαδικασία, Τέλος, ε, πιστεύω πως η διαδικασία θα γίνει πιο διάφανη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση και πρέπει να τη χειριστούμε με όσο το δυνατόν ε, πιο διάφανο και δημοκρατικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να αλλάξει η διαδικασία και να μην δοθεί η εντολή για τις διαπραγματεύσεις τώρα, αλλά να περιμένουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρέπει να πω πως δεν συμφωνώ μαζί σας για ε, τα όσα είπατε περί διαφάνειας και δημοκρατικότητας, διότι ακολουθούμε ακριβώς τον πιο δημοκρατικό και ε, διάφανο ε, τρόπο λειτουργίας για το θέμα αυτό. Ενημερωνόμαστε για όλες τις συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών, συμμετέχουν όλοι οι εισηγητές και οι σκιώδες εισηγητές των άλλων επιτροπών και μπορώ να πω πως η διαφάνεια είναι δεδομένη. Εσείς προτείνετε να λάβουμε εντολή από την Ολομέλεια, δηλαδή να γίνει η πρώτη ανάγνωση και εντολή από την Ολομέλεια. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τους συνεισηγητές εάν συμφωνούν τι άποψη έχουν. Πρόκειται για μία πρόταση αλλαγή της διαδικασίας στο τέλος αυτής εδώ της διαδικασίας. Εσείς ως συνεισηγητές είχατε την ευκαιρία να το συζητήσετε κατά τις συνεδριάσεις των ε, Βρισκόμαστε δύο βήματα πριν το τέλος, πριν τις διαπραγματεύσεις, πριν την Ολομέλεια και εσείς προτείνετε αλλαγή. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη των συνεισυχητών. Κύριε Βανίστελ Ρόι. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ, αλλά διαφωνούμε. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων με τους ε, σκιώδεις εισηγητές, αλλά και με τους εκπροσώπους των άλλων επιτροπών, ετέθη το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και υπήρχε μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία επιθυμούσε να ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας και να μην περάσουμε στην ελομέλεια. Και υποθέτω πως είστε κατά Τη όλη πρόταση εν γέννη, γι' αυτό προσπαθείτε να υπονομεύσετε το αποτέλεσμα με αυτήν την πρόταση. Νομίζω ότι η πρότασή σας δεν έγινε δεκτή ούτε από την πλειοψηφία των σκιωδών, ούτε από τους εκπροσώπους των άλλων επιτροπών. Αυτό έχω να πω ως απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα και με τους δυο σας. Οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια με όλες τις ε, συνδεδεμένες επιτροπές, με όλους τους κοιόδης. Ε, πιστεύω πως έχουμε αρκετά μεγάλη δύναμη για να προχωρήσουμε μόνοι μας στον τριμερή διάλογο και θεωρώ πως εμείς ως Επιτροπή ε, χαρακτηριζόμαστε από διαφάνεια και από νομιμότητα. Γι' αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ανέφερα, Σήμερα έχουμε τρεις ψηφοφορίες στο τέλος του καταλόγου ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες, θα ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση και στο τέλος θα ψηφίσουμε την διαπραγματευτική εντολή. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας η Επιτροπή δεν συμφωνήσει να δώσει εντολή, αυτό θα σημαίνει ότι Όλη η Επιτροπή στηρίζει εσάς. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την υφιστάμενη διαδικασία. Να σας υπενθυμίσω πως ε, σχεδόν ένα χρόνο ε, ασχολούμαστε με αυτό και προτείνω να αρχίσουμε αμέσως. Όπως και να έχει θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Με συγχωρείτε προ διευκρίνηση, κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το διαδικαστικό σημείο τώρα και μετά να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία ανάλογα με το αποτέλεσμα τη ε, ψηφοφορία που προτείνω. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία με λεπτομέρειες, αλλά, θα, αλλά αυτό ζητώ να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Αν υπάρχει πλειοψηφία που επιθυμεί να συνεχίσουμε με την ε, διαδικασία που προτείνω, να την ακολουθήσουμε και αν όχι, να ακολουθήσουμε τον εσωτερικό κανονισμό, έτσι όπως έχουμε αρχίσει. Είναι μια πρόταση αυτή μόνο. Η κυρία Κρέλ, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Ο κανονισμός ε, αναφέρει ότι πρώτα ψηφίζουμε την ε, πρόταση των εισηγητών. Όλα τα χρόνια που είμαι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έτσι κάνουμε. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν. Έχουμε ψηφοφορία. Πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση τις τροπολογίες των εισηγητών, το συμβιβαστικό κείμενο και στο τέλος όλων αυτών θα ψηφίσουμε για το αν θέλουμε να δώσουμε εντολή στην πρόεδρο, τους ε, συνεισηγητές, τους κοιόδες εισηγητές και τους εισηγητές των άλλων επιτροπών να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Και αυτή είναι η στιγμή όπου θα κληθούν τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν. Αρχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία για τις τροπολογίες. Okay. We do not... Δεν ψηφίζουμε λοιπόν την πρώτη τροπολογία, την 59. Έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 60 λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Έκον 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έκον 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλτ 14. με Επιτροπή Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 5. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 νέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 247. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πες τρία, Αλία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 249. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εμπλή 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κρίνεται. 258. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζ 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Μπάτζ 13. Το βρήκατε. Επαναλαμβάνω. Μπάτζε 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 260. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Budget 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλο 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλο 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλο 85. Όχι, η έμπλο 85 καταπίπτει γιατί απορρίφθηκαν οι προηγούμενε τροπολογίες. Θα περάσουμε τώρα στην τροπολογία 200. Όχι. «261. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 262. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλτ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 1 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Έκον 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10 καταπίπτει και θα περάσουμε στη συμβιβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εμπλυ 12. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Budget 2. Τη βρήκατε όλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κάλτ 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Όχι, με συγχωρείτε. Τροπολογία 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ας το κάνουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 125 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πες 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1. Ε, θέλετε να τοποθετηθείτε γι' αυτή, όχι. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 1 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Πρώτη από τις τελικές ψηφοφορίες, τελική ψηφοφορία για το σύνολο των τροπολογιών. Η ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Βλέπετε κι εσείς. Ναι. Τελευταία ψηφοφορία ψηφίζουμε για, τις, για την εντολή για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων, σύσταση διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως γνωρίζετε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 29 ψήφοι πέρα, 11 κατά. Συγχαρητήρια στους εισηγητές. Okay, now we continue with, um, um, Και τώρα περνάμε στην έκθεση του κυρίου Βανίστε Ρόι επενδύοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση βελτιστοποίηση της συμβολής Ευρωπαϊκών Διαθροντικών και Επενδυτικών Ταμείων αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο υπαριθμών 16. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Βανίστερο. Όχι. Εντάξει. Ξεκινάμε με τον συμβασμό υπερθμών 1. Πέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική υπερθμών 2. Ψήφι πέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθμών 4. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία υπερθμών 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή Σύμβαση, ε, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 7 σε, δύο, σε 3 τμήματα συγγνώμη πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική πρόταση υπερθμών 8. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική 9. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική 10 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ με τις κάρτες σας. Ψηφίζουμε τροπολογία 110 ηλεκτρονικός αρχιτεκτό ψηφοφορία. Πέρας αυτής απορρίφτεται. Τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίπερ κατά αποχές λεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απο... Ε, δεκτό. Τροπολογία 121 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να επαληθεύσουμε επαλήθευση επί της 121 ψηφίζουμε η ψηφορία The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας ε, έχει απορριφθεί. 122 τροπολογία ψήφι πέρα. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 16 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, συγγνώμη εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτό Τροπολογία 143. Υπέρ, κατά, αποχές, ας επαληθεύσουμε. Τροπολογία 123, ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς, Άρχιτε ψηφοφορία. The vote is closed. η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρί. Θέλετε επαλήθευση. Mm. Ωραία. Επαληθεύουμε. Τροπολογία 181. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς. Άρχιτη ψηφορία. The vote is closed. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Αρχικό κείμενο. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία υπερθμών 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 25 υπέρ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 196 τροπολογία υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε 196 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώ. The vote is closed. Η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 197 τροπολογία ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία, ε, ε συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 207 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 208 τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθυμό 29 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 227 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 239 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 240 υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεκτή. Τροπολογία 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία του προπολογισμού 2 ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 246 τροπολογία. 47 συγγνώμη. Ψήφι υπέρ της 247. Κατά αποχές δεκτή. 249 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία υπαρθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προλογία 2 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Προλογία 3 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίθηκε. Προλογία 4 υπέρ, κατά, εποχές, νομίζω πως έχει απορριφθεί, αλλά σε επαληθεύσουμε. Προπολογία 4, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικός, αρχή ψηφοφορία. πέρας έχει απορριφθεί. Συμβαστική 34. Ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εκτιμώντας C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά, ε, εγκρίθηκε. Συμβαστική 35, 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε. Ας επαληθεύσουμε. Τροπολογία υπερθυμών 21 ηλεκτρονικός παρακαλώ. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή εγώ έσφαλα, συγγνώμη. Τροπολογία 40. Συμβαστική. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 36. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 37. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προπολογία 33 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απερίφθη. Προπολογία 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 39 υπέρ κατά εποχές δεκτή. Περνάμε στην ε, employment απασχόληση υπάρχουν 7. Ναι, υπάρχει μόνο 7 της επιστήμης απασχόλησης. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Θέλετε επαλήθευση επί τις 7. Θα ελέγξουμε. Άρχη ψηφορία. Έληξε και έχει γίνει δεκτή. 9 έμπλ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην τρέν 7 ψήφι κατά αποχές δεκτή. Τρέν 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άγκρι 21 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απερίφθη αλλά σε επαληθέψουμε. άγκρι υπερθμών 21 ψηφίζουμε ηλεκτρονικός άρχιτε ψηφοφορία The vote is απορρίφθηκε. Περνάμε στην συμβαστική. Συγγνώμη, έχουμε την άγρη 30 ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβαστική 41 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καλτ 21 υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές δεκτή. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρα ψηφοφορίας και η έκθεση έγινε δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Βανίστα Ρόι. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. We go to the next vote. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση. Ο κύριος Νίλσον είναι ο συντάκτης γνωμοδότησής μας. Ξεκινούμε με τη συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κα... Συγγνώμη, συγγνώμη. Γιατί είναι 8 μιλάω. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 8. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια κύριε Νίλσον. Νίλσον. Νίλσον. Εδώ ολοκληρώνεται η ψηφοφορία μας. Συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για έκθεση πρωτοβουλίας μελλοντικές προοπτικές τεχνικής αρρωγής για την πολιτική συνοχής. Μισό λεπτό. Okay, can we continue now? Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. I think we can. Νομίζω ότι μπορούμε. Λοιπόν, πρώτη εντελεγή απόψεων για την έκθεση πρωτοβουλίας για τις μελλοντικέ προοπτικές τεχνικής αρρωγής για την πολιτική συνοχής. Ο εισηγητής μας, Ρούζα Τόμασιτς, η εισηγητριά μας, συγγνώμη, θα μας ε, κάνει μια πρώτη παρουσίαση της δουλειάς της. Ε, ευχαριστώ πολύ, παρά το γεγονός ότι η τεχνική αρρωγή έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής από το 1988. Μια σφαιρική ανάλυση συμμετοχής της και του ρόλου της δεν έχει γίνει ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η τεχνική αρρωγή είναι ένα βασικό στοιχείο δαπανών για το οποίο δεν υπάρχει κανένα σαφής ορισμός. Είναι δύσκολο να γίνει λεπτομερής αξιολόγηση της σημασίας της και της συμμετοχής της στην ενίσχυση ε, των, ε, των θεσμών, όπως επίσης και την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας για τα επενδυτικά κονδύλια. Και επειδή μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές δημοσιονομικές γραμμές και είναι δύσκολη η ευέλικτη χρήση Είναι δύσκολο να ξέρουμε τα τελικά ποσά ή ε, να έχουμε μια σαφή κατανόηση των, ε, ε, ε, ε δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί είχαν υπάρξει κατά την τελευταία προγραμματική περίοδο ε, κάποιες αλλαγές που αφορούν κυρίως την ε, διοικητική ανάπτυξη ικανότητας και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας με σκοπό να τεθούν προτεραιότητες και να εφαρμοστούν διοικητικές ε, μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις σε κάποια κράτη-μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 100 18 του κοινού ε, κανονισμού, του, κανονισμού κοινών διατάξεων αυτή τη στιγμή έχουμε 0,35% ε, ε, των ποσών αυτών ως τμήμα του συνολικού προπολογισμού αύξηση 0,1% σε σχέση με την περίοδο 2010-2013. Μεταξύ άλλων, η τεχνική αρρωγή υποστηρίζει την ενίσχυση των θεσμών και της διοικητική ικανότητα για την καλή διαχείριση των κονδυλίων. Θα ήθελα να πω ότι με χαρά αναγνωρίζω τις δύο τελευταίες εξελίξεις ε, με ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ικανοτήτων ε, όπως επίσης και ένα μηχανισμό ε, εξασφάλισης των ενωσιακών κονδυλίων. Υπάρχει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση του ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ το άλλο εργαλείο είναι προσαρμόσιμο με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες δομές των κρατών μελών. Το πιλωτικό πρόγραμμα, ε, το σύμφωνο Ακεραιότητας για την ε, εξασφάλιση των κονδυλίων ε, έχει σκοπό τη διασφάλιση των κονδυλίων κατά της διαφθοράς και της απάτης με σκοπό την ανάπτυξη της λογοδοσίας, την ενίσχυση των, αρμοδιών, των αρμοδίων αρχών κατά την σύναψη συμβάσεων με καλύτερο ανταγωνισμό ε, και ε, καλύτερες δημόσιες προμήθειες. Σε επίπεδο κρατών μελών μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια περίπου. Ε, ευρώ, η τεχνική αρρωγή μπορεί να θεωρηθεί ε, ως μοχλός αλλαγής και τα πλήρη ωφέλη της είναι εμφανή ε, στο μέλλον όταν οι δραστηριότητες και οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν πλήρως ολοκληρωθεί. Επομένως, ε, η διαφάνεια των δραστηριοτήτων τεχνικής αρρωγής πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε ε, στάδιο. Η σημασία της ε, για τη θεσμική και διοικητική μεταρρύθμιση στα κράτη-μέλη πρέπει να γίνεται σωστά ώστε να υπάρχει νομιμότητα και λογοδοσία. Όσον αφορά την ενίσχυση των θεσμών και της διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών, η χρήση των κονδυλίων ποτέ ε, δεν έχει γίνει σε ε, τοπική περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δηλαδή έχουν χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο ε, για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ φορέων που δεν μπόρεσαν όμως να εκφράσουν τις ανάγκες τους γιατί δεν υπήρχε καμία προσπάθεια ε, συμπερίληψης της άποψής τους, ούτε ως προς την κατάργηση. Ελπίζουμε λοιπόν να, να βελτιώσουμε την τεχνική αρρωγή για τα επόμενα έτη, γιατί ο σκοπός της δεν είναι απλώς να ξοδεύονται χρήματα, αλλά να χρησιμοποιούνται για στοχευμένες ομάδες συμμετεχόντων, να ενημερώνονται η τοπική και περιφερειακή περιφερειακοί σε γέρο για όλε τι δυνατότητε τεχνική αρρωγή, ώστε η κατάρτιση, η οποία οργανώνεται από τα κράτη-μέλη, να μπορεί πράγματι να δημιουργήσει μια προστιθέμενη αξία προ προς τις ανάγκες που υπάρχουν και να γίνεται και μια καλή αξιολόγησή τη από του συμμετέχοντες. Επίση, πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε στο πλαίσιο τη τρέχουσα ατζέντα ε, τη αστική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει τέτοιου είδου αρρωγή για όλε τι δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία δημιουργία του συστήματος, όπως επίσης και με την εφαρμογή των έργων ε, σε ολόκληρη την επικράτεια, γιατί οι πόλεις γίνονται ενδιάμεση φορείς ε, στην ε, αξιολόγηση και την εφαρμογή των προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη τεχνική αρρωγή και οι σχετικέ διευκολύνσει ε, εφαρμόζονται επιτυχώ σε κάποια κράτη-μέλη. Ωστόσο, περισσότερε πληροφορίε για τι ευκαιρίε αυτές ε, χρειάζονται και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Ένα σημαντικό ε, συντελεστή επιτυχία είναι η ευαισθητοποίηση για κάθε πρόγραμμα. Πρέπει να υπάρχουν σαφεί επεξηγήσει για τους υποψηφίου, να γνωρίζουν την τεχνική αρρωγή και η κρίση στην Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει να έχει υπάρχει μια ευελιξία στα διαρθρωτικά και τα επενδυτικά ταμεία, κάτι το οποίο αντανακλάται στις ε, διατάξεις που αφορούν ε, την τεχνική αρρωγή. Το άρθρο 25 του κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις μπορεί να ισχύει στα κράτη-μέλη με προσωρινές οικονομικές δυσκολίες, όμως μια πιθανή επέκταση του γεωγραφικού, ε, της γεωγραφικής εμβέλειας συζητείται αυτή τη στιγμή ε, στο πλαίσιο μια νέας νομοθετικής ε, πρότασης το πρόγραμμα ε, ενίσχυσης των διαθετικών αλλαγών πρέπει να είναι συμπληρωματικό για της τεχνικής αρρωγής ε, υπό τα ενωσιακά διαθροτικά και επενδυτικά ταμεία. Πώς μπορούμε όμως να εξασφαλίσουμε την σχέση μεταξύ ε, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμματισμένων δράσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Χρειάζεται λοιπόν περισσότεροι πόροι που θα είναι στη διάθεση των κρατών μελών. Ε, η κατανομή των δραστηριοτήτων τεχνικής αρωτη... Ε, τεχνικής αρρωγής πρέπει να γίνεται καλύτερα και πιο στοιχειοθετημένα ε, το, ε, προβλέπεται ένα σχετικό σεμινάριο για το 2017 και την ίδια μέρα θα γίνει μια συζήτηση και στην ε, Επιτροπή μας για το θέμα αυτό με, την, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα λεπτομερώς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Μας ενημερώσατε για την ημερομηνία παρουσίασης του σχεδίου έκθεσης. Εμείς θα συζητήσουμε τι τροπολογίε, θα αποφασίσουμε σχετικά και θα συνεχίσουμε. Ψηφοφορία λοιπόν είναι προγραμματισμένη για το Μάρτιο του 2017 και τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδει εισηγητές. Κύριε Σπυράκη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τα σχόλια της κυρίας Τόμασιτς και να πω πως ε, θα ήθελα να παραμείνει αυτός ο σαφής ε, ορισμός του πώς θα εισάγεται η τεχνική βοήθεια, η ανάγκη για διαφάνεια και η ανάγκη για αποτελέσματα. Τα 10 δισεκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και να πω δύο λόγια ε, συμπληρωματικά σε αυτά που είπε η κυρία Τόμασιτς το πρόγραμμα στήριξη διαθροτικών μεταρρυθμίσεων είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα έχει επιπτώσει στο μέλλον τη τεχνική βοήθεια και πρέπει σίγουρα να ληφθεί υπόψη σε όλες τις σχετικές συζητήσει. Φυσικά στη συζήτηση πρέπει να ε, εισαγάγουμε και πρακτικές λύσεις και να σας δώσω ένα παράδειγμα της χώρας μου. Η Task Force για την Ελλάδα ε, και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου για ε, αυτό πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά και το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού Περικοινών Διατάξεων η Ελλάδα έλαβε ε, χρηματική βοήθεια για τεχνική στήριξη αλλά δεν είδε αποτελέσματα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψή μου, επομένως, χρειάζονται προσαρμοσμένα όργανα τα οποία θα έχουν και ευελιξία δημοσιονομική. Χρειάζεται η κατάλληλη τεχνική βοήθεια κατόπιν ε, ζήτησης. Γι' αυτό λοιπόν θα χαρώ να συζητήσω με τους συναδέλφους μου για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τόμασιτς και α, θα συνεργαστούμε, είμαι σίγουρη, πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέλ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του σκιώδου συγγητή κ. Κοσολίνο. Έπρεπε να φύγει γιατί προέκυψε κάτι και δεν είμαι ε, καλά προετοιμασμένη για να τον αντικαταστήσω. Θα ήθελα όμως να ζητήσω, να παρακαλέσω την ε, η συγγήτρια να συμπεριλάβει και τα ακόλουθα σημεία στο σχέδιο έκθεσης. Καταρχάς, ο, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για την τεχνική βοήθεια. Αυτό ήταν αναγκαίο. Δεν υπήρξε διαφωνία γι' αυτό. Όμως, εδώ το ζητούμενο είναι ε, τι γίνεται με τις ε, συνεργασίες, με την αρχή τη, των, ε, της ε, με τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και πώς αυτό θα συνδεθεί με την πολιτική συνοχή. Αυτό όλο πρέπει να συζητηθεί, να δούμε και τι γίνεται με τη διοικητική ικανότητα, με το πώς θα διαχειριστούμε τα ταμεία. Αυτό είναι κάτι που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι το οποίο ούτε τα κρατημέλη ούτε οι Κομισιόν έδειξαν προθυμία να ε, συζητήσουν, να προχωρήσουν. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνική βοήθεια με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε δει εκπληκτικά αποτελέσματα βελτίωση της διοίκηση ε, που ωφελούν τους νέους ανθρώπους, που βοηθούν ε, την ε, χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Ίσως λοιπόν καταφέρουμε να βρούμε μια δυνατότητα όταν διατίθεται δημόσιο χρήμα, για παράδειγμα, για την ε, κατάρτιση των ε, διοικητικών υπαλλήλων. Να βοηθάει αυτό όχι μόνο ε, τους ίδιους τους υπαλλήλους, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και να έχει ευρύτερες, θετικότερες συνέπειες στην πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέλ. Εγώ είμαι η επόμενη σκιώδη εισηγήτρια. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω δύο λόγια. Να πω καταρχά συγχαρητήρια για τις ε, ιδέες αυτές, τις προτάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια αξιολόγηση και κατόπιν να στηρίξουμε την τεχνική βοήθεια για την πολιτική συνοχή. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις ε, από πολλές πτυχές, οικονομικές, ε, και τα λοιπά. Υπάρχει επίσης και το θέμα της προστιθέμενης αξίας της τεχνικής βοήθειας. Διότι είναι ένα στο κομμάτι της πολιτικής συνοχής και πρέπει να βρούμε προστιθέμενη αξία σε κάθε ένα από τα στάδια της τεχνικής ε, βοήθειας. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν δείκτες για σχεδόν όλες τις δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων αλλά σπάνια υπάρχουν δείκτες για την τεχνική βοήθεια και την επιτυχία της. Ε, είτε σε εθνικό επίπεδο, μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων είτε αλλιώ. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω απόλυτα την προσπάθεια που κάνετε για να μετρηθεί η προστιθέμενη αξία της τεχνικής βοήθειας. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διεθνωτικά ταμεία, αλλά και διότι η τεχνική βοήθεια συμπεριλαμβάνει όλους τους δικαιούχους, όλους τους αρμόδιους φορείς, ε, τους, ε, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις επιτροπές παρακολούθησης, ε, συμπεριλαμβάνει όλα τα στάδια της εφαρμογής ενός προγράμματος, της χρήσης των διορθωτικών ταμείων. Θα επιθυμούσα στην έκθεση να συμπεριληφθεί και ο ρόλος της τεχνικής βοήθειας στην εδαφική συνεργασία, για την εδαφική συνοχή στα προγράμματα για διασυνοριακή συνεργασία, διεθνή, διεθνική συνεργασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό η τεχνική βοήθεια να χρησιμοποιείται ε, με τρόπο χρηστό για προσπάθειες κοινέ, έτσι ώστε να δοθεί ακόμα υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Αυτό χαρακτηρίζει την επιτυχία ενός προγράμματος. Συμφωνώ απόλυτα ότι η τεχνική βοήθεια πρέπει να είναι ένα ευέλικτο μέσο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα για να στηρίξουμε τα κρατημέλη στην προσπάθειά τους να μεταρρυθμίσουν τη διοίκησή τους και άλλους στρατηγικούς τομείς. Και σίγουρα η δική σας έκθεση και η έκθεση νομοθετικού περιεχομένου που μόλις ψηφίσαμε σχετίζονται. Γι' αυτό λοιπόν θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί σας ως και ηγήτρια για την έκθεση αυτή και θα σας στηρίξω στις προσπάθειες και στην σκληρή δουλειά που σίγουρα θα κάνετε. Ε, ο επόμενος σκιώδης εισηγητής, όχι δεν έχουμε. Κύριε Μάτο, εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αδικαστώ και εγώ τη συνάδελφο. Γνωρίζουμε πως μία από τις χρόνιες προβληματικές της πολιτικής συνοχής αφορά τις διοικητικές ικανότητες. Δεν αποτελεί μυστήριο το ότι ε, μία συμμετοχή σε, αυτά τα, σε αυτές τα προγράμματα αποτελεί πρόκληση για τις τοπικές αρχές. Συχνά πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες ε, δεν μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν την νομοθεσία και τους κανονισμούς τηρώντας το Σύμφωνο Σταθερότητας και το 2014 τηρώντας ε, την, ε, τη μακροοικονομική ε, ρεσιμότητα. Είναι καλό λοιπόν στον ισχύοντα κανονισμό να προβλεφθούν μέτρα τα οποία θα στηρίζουν τις άμεσες δράσεις για να περιορίσουν τα διοικητικό κόστος και να βελτιώσουν την χρησιμοποίηση των, των πόρων των δικαιούχων. Όπως επίσης είναι καλό να προαχθούν οι επενδύσεις ε, από τις αρχές και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών και αυτό σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης και σε τούτου να υπάρξει ένα ε, θεσμικό πλαίσιο πιο αποτελεσματικό για να υπάρξει καλύτερη διακυβέρνηση. Θα ήθελα να εκφράσω όμως κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την πιθανή ε, σχετισμό με τα διαφορετικά προγράμματα. Τα, τα χρήματα υπάρχουν. Μιλάμε για το θεματικό 11, περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, 6,5 με την εθνική συγχρηματοδότηση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου που έχει ένα πρόγραμμα 827 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως αυτοί οι πόροι να μην χρησιμοποιούνται με τρόπο ορθό. Χρειάζεται άρα να ελέγξουμε το πώς δαπανώνται ή θα ε, παρακάψουμε τα προγράμματα αυτά και ε, δεν θα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ενορχιστρωμένο από έναν ε, επίτροπο που έχει ως στόχο τη μείωση των πόρων αυτών της συνοχής. Συχνά το ξεχνάμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει περιμένω την ε, αντίδραση της συναδέλφου, την οποία ευχαριστώ για το σημαντικό θέμα που την απασχόλησε. you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοφτσετς έχει τη στο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τόμασιτς για την έκθεσή του στην οποία βλέπουμε αρκετά ενδιαφέρουσες ε, υποθέσεις και προτάσεις. Αλλά θα ήθελα να, μιλήσω από προσωπική εμπειρία. Για 12 χρόνια ε, προείδρευσα μιας εδαφικής περιφέρειας ε, την Ζουπάνη στην Κροατία. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά τι σημαίνει τεχνική αρρωγή. Ε, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να χορηγείται αυτή η τεχνική αρρωγή πιο εύκολα και να είναι πιο διαθέσιμη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, όπως και αν τις ονομάζουμε στα διάφορα κρατημέλη. Και αυτό περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή. Εξάλλου, ε, σημασία έχει να επιτρέψουμε την διασυνοριακή τεχνική αρρωγή, διότι υπάρχουν μια σειρά από διασυνοριακά προγράμματα, τα, τα οποία δεν ε, επιτυχάνουν διότι δεν υπάρχει αρκετή γνώση, τεχνογνωσία, ικανότητες και από τις δύο πλευρές. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κυρία Τόμασέτσου για τις προτάσεις και τις συστάσεις. Ευχαριστώ. Μια που δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Επευθύνομαι στους εκπροσώπους της Κομισιόν. Ποιος θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνει το λόγο. Είμαι επικεφαλής ε, της μονάδας που ασχολείται με το ζήτημα των, ε, της τεχνικής βοήθειας ε, στην DG Regio. Να σας πω φυσικά ότι είναι πρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και προσβλέπουμε τα συμπεράσματα της εκθέσεώς σας, να δούμε πώς μπορούν να συμπεριληφθούν στις εργασίες μας. Έχουμε μία συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο για να κάνουμε ανταλλαγή των απόψεών μας. Όταν μιλάμε για τεχνική αρρωγή, φυσικά υπάρχει εσωτερική τεχνική αρρωγή με την πρωτοβουλία της Κομισιόν, η οποία είναι σημαντική, αλλά είναι πολύ χαμηλότερη από τα τεχνικά αρρωγή που παρέχεται από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τεχνική αρρωγή που είναι η από εμάς Κομισιόν. Έχουμε ήδη παρακολουθήσει εδώ και αρκετά χρόνια μια στρατηγική προσέγγιση για το πώς θα χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική αρρωγή και έχουμε αναπτύξει μια εσωτερική στρατηγική που, αφορά, που περιέχει έξι προτεραιότητε. Η μονάδα μα είναι επικεφαλή στα θέματα που αφορούν την ε, διοικητική ικανότητα και την οικοδόμηση. Παίζει τα πακέτα ολοκλήρωση ε, μεταξύ ομοτήμων, όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την τεχνική αρρωγή για τα οποία ασχολείται η μονάδα μα. Έχουμε επικεντρώσει ε, σε πέντε στοχείς σε πέντε τομείς, ε, επικαιροποίηση, την καταπολέμηση της ε, απάτης, ε, ανταλλαγή βρίσκων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και περιφέρειες. Αυτή λοιπόν είναι η στόχη μας όπου αναπτύσσουμε νέες πρωτοβουλίες και νέες αναλύσεις. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες χρειάζονται. Τώρα, για τα επιχειρησιακά προγράμματα, το ποσό ανέρχεται σε 10 δις ευρώ για διαβολεύσεις 2014-2020 ακολουθούμε μια προσέγγιση που ζητάμε τα κρατημέλη να κεντρώσουν ιδιαίτερα στα ζητήματα κλειδί που τα απασχολούν. Έχουμε ήδη εμπλακεί σημαντικά στον προγραμματισμό αυτών των ε, τεχνικών ε, τεχνικής βοήθειας και η βοήθεια φυσικά αφορά την χρηματοδότηση κατάρτισης ε, ανθρωπίνου δυναμικού και υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης παρόμοιου δυναμικού για να αρχίσουν να προσλαμβάνουν νέα πρόσωπα, νέα άτομα. Αυτό φυσικά απαιτείται ακόμη περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε ενδιάμεσους οργανισμούς. Οι προσλήψεις φυσικά θα γίνουν σε, στο κράτος μέλος. Υπάρχει και το ζήτημα της τεχνικής αρρωγής για το θέμα της ε, ε, εκ των υστέρων αιρεσιμότητας ε, και έχουμε επιφυλάξει, έχουμε κρατήσει χρήματα για την καταπολέμηση των διαφθοράσεων. Ε, προσπαθούμε ήδη να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική αρρωγή πολύ περισσότερο με στοχευμένο και εστιασμένο τρόπο. Όταν μιλάμε για δείκτες, ε, οι δείκτες είναι ακόμα αρκετά αδύναμοι σε θέματα τεχνικής βοήθειας, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες ε, πληροφορίες για το τι προσωπικό απαιτείται για αυτή την τεχνική αρρωγή κλπ. Θα λάβουμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες πάνω στα θέματα αυτά, πόσες ε, θέσεις θα χρηματοδοτήσουμε για θέματα τεχνικής βοήθειας. Σας είπα ότι προσβλέπουμε στα συμπεράσματά σας και με τα χαρά θα συμμετάσχουμε στο εργαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, πολύ σύντομη θα είμαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συμβολή τους. Τα σημείωσα όλα, όλες τους τις προτάσεις και ελπίζω ότι θα με βοηθήσουν ε, να συντάξω την καλύτερη έκθεση που έχει συνταχθεί ποτέ. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας. ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την απαλλαγή 2015 ε, Γενικός προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, αυτή τη στιγμή εξετάζει την απαλλαγή του 2015 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μας γνωμοδοτεί και εγώ είμαι η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Ε, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε το πρόγραμμά μας με την Αρμόδια Επιτροπή πρέπει να ψηφίσουμε στις 24 Ιανουαρίου την γνωμοδότησή μας ε, του 2017. Οι σκιώδεις ηγητές χρειάζονται χρόνο για να εξετάσουν τις τροπολογίες, οπότε προτείνω μία προθεσμία τροπολογιών 12 το μεσημέρι στις 12 Δεκεμβρίου. 12 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Θα ήθελα τώρα να σας πω ποια είναι η άποψή μου για την γνωμοδότηση που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά θα σας τα πω στα βουλγαρικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζουμε όλοι, η διαδικασία της απαλλαγής είναι μία ευκαιρία να εκφράσουμε την άποψη της Επιτροπής μας ε, όσον αφορά την εκπλήρωση της ετήσιας ε, ε, έκθεσης του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας παρουσιάζω τα βασικά στοιχεία της γνωμοδότησης. Το 2015 σημειώνουμε ότι το επίπεδο των σφαλμάτων έχει μειωθεί από 5,6 του 2014 σε 5,2% για το 2015 το οποίο είναι αποτέλεσμα βέβαια της βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ε, από τα κράτη-μέλη και των συλλογικών μέτρων που ε, υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικές πηγές των σφαλμάτων ε, εντοπίστηκαν κατά τη χρήση κανόνων που αφορούσαν την, τις κρατικές ενισχύσεις και τη λογοδοσία το, το 2015, ε, τα σφάλματα του 2015 μπορούν να διορθωθούν πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσέξει όλος ιδιαίτερος ε, ε, όσον αφορά το παραδεκτό κάποιων κανόνων των κρατών μελών σε σχέση με το ΦΠΑ και να δοθεί να δοθούν ε, σωστές οδηγίες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι τα κράτη-μέλη ε, παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα αναχρηματοδότησης για το 2015 σε σχέση με το 2014, κάτι το οποίο είχε αποτέλεσμα της μείωσης του επίπεδου των ε, μη επιστροφών σε σχέση με το 2015 και επίσης καλύφθηκαν αρκετές καθυστερήσεις όσον αφορά την ε, εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο, νομίζουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ε, αυξημένος ε, καθυστέρησης εκτέλεσης προϋπολογισμού την επόμενη χρονιά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το τέλος του 2015 είχαμε διαπιστώσει ε, ότι 10% ε, των κρατικών φορέων ε, ε, καθυστερούσαν ε, και είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει και να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Στις 30 Ιουνίου 2016 οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες των κρατών μελών δεν είχαν ακόμη μεταγραφεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τα κράτη-μέλη στην εκτέλεση των σχεδίων δράσης τους ε, που βασίζονταν βέβαια σε, προηγούμενες, ε, σε προηγούμενους κανόνες. 1025 ε, οι οικονομικά εργαλεία ε, χρησιμοποιήθηκαν, οικονομικά μέσα, 10% αύξηση σε σχέση με το 2013. Επίσης γνωρίζουμε και το θέμα του λογιστικού ελέγχου σε σχέση με την παράταση της ε, προθεσμίας για να λάβουν τα κονδύλια οι τελικοί χρήστες μέσω απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντί τροποποίησης του κανονισμού. Γιατί αυτό μπορεί μπορούσε να συμβεί μετά την 30 Δεκεμβρίου του 2015 μόνο. Επίσης η γνωμοδότηση σημειώνει τις προτάσεις για την εκ νέου ε, αξιολόγηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τη μεγαλύτερη ευελιξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και όλα τα, κράτη και όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης καλούνται, για, καλούνται να αναθεωρήσουν τη δομή των ε, επενδυτικών ταμείων. Μέχρι το 2020 πρέπει να λάβουν υπόψη την άποψη της ομάδας υψηλού επίπεδου. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι Συμφωνώ με την άποψη ε, της ελεγκτικής υπηρεσίας, ότι δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε όλα τα αποτελέσματα που προσμετρούν τη συνεισφορά όλων των εταίρων στην επίτευξη των στόχων. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την σύντομη παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης ηγητές. Κύριε Πότσακ, έχετε το λόγο. Όχι, λάθος όνομα είπατε, δεν είμαι εγώ αυτός. Είναι λάθος η σειρά. Σωστό το όνομα, λάθος η σειρά. Θα μιλήσετε μετά. Ξέρω πως ε, μπορώ να επινοήσω όποιο όνομα θέλω και εσείς να το δεχτείτε. Αυτή τη φορά όμως δεν έκανα λάθος. Έχετε το λόγο κύριε Πόλτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την έκθεση απαλλαγή το 2015. Η γνωμοδότηση αυτή είναι, θεωρώ, ένας καλός απολογισμός ε, της κατάστασης. Ε, φαίνονται οι προκλήσεις, οι καθυστερήσεις δηλαδή της προγραμματικής περίοδου, από το 2014 στο 2020 που ακούσαμε και νωρίτερα από την κυρία Πίτροπο η οποία μας εξέθεσε τη δική της άποψη. Επίσης, η ελλείψη στην υλοποίηση της οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες ή ο χαμηλός όγκος αποζημιώσεων από τις αρχές, τις αρχές. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε κάποιες τροπολογίες της νομοδότησης. Βλέπω ότι ο αριθμός των σφαλμάτων έχει μειωθεί από τα προηγούμενα έτη. Αυτό φαίνεται αρχικά θετικό. Όμως ε, τα ποσοστά αυτά είναι στα ίδια επίπεδα του 2014. Κάτι που θεωρώ πως δεν είναι τόσο καλό. Σε σχέση με την απαλλαγή του 2014, στη γνωμοδότηση μου λείπουν κάποια σχόλια, ότι δηλαδή δεν είναι όλες οι παρατυπίες αποτέλεσμα απάτης. Πολλές φορές οφείλονται σε έλλειψη πληροφόρησης, γνώσης, σε, κάποιες, ε, σε κάποια μικροπροβλήματα σχετικά με το νομικό πλαίσιο. Και νομίζω πως αυτό πρέπει να αναφερθεί ακριβώς δεδομένης της εικόνας που έχει η περιφερειακή πολιτική, διότι ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει αυτή την έκθεση και να σταθεί μόνο στην ε, απάτη. Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εντυπώσεις. Αυτό που μου λείπει επίσης από την έκθεση είναι κάποια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη και στους αρμόδιους φορείς να διασφαλίσουν πως οι δικαιούχοι των Ευρωπαϊκών Ταμείων θα είναι ενημερωμένοι για τις προϋποθέσεις άντλησης κονδυλίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι υποχρέωση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση και μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και θα ε, δούμε βέβαια τι θα γίνει στην ψηφοφορία και γι' αυτό λοιπόν ε, θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Έχετε τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Προφέρετε το όνομά μου σωστά. Βον. Έτσι ονομάζομαι. Λοιπόν, Βλέπω με πολύ θετικό μάτι το ότι υπάρχει μείωση στον αριθμό των σφαλμάτων, ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις ε, ως προς τον έλεγχο της διαχείρισης, ως προς τις διορθώσεις. Πιστεύω ότι οι λόγοι για τα σφάλματα δεν είναι άγνωστοι, όπως είπατε κι εσείς, είναι γνωστοί. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες επιλεξιμότητας για τις δημόσιες προμήθειες, και ακριβώ εξαιτία όλων αυτών θεωρώ πω είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει κάποια ε, πρόοδο στην ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου. Πρέπει να δούμε πρόοδο εκεί για να δούμε και ποιες είναι οι συστάσεις τους, να δούμε πώς μπορούμε να τις ε, εφαρμόσουμε. Όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίσαμε και αυτήν την ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου. Επίσης, να πω πως αξίζει να σημειωθεί ο ρόλος των κρατών μελών εδώ στην απλούστευση. Για παράδειγμα, τα ίδια τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ε, μειώσουν τα ίδια τη γραφειοκρατία στο μέλλον, να υποβάλουν κάποια μελέτη, κάποια ανάλυση του προβλήματος και όσον αφορά τις ε, δημοσίες προμήθειες είπατε κι εσείς ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν μεταφέρει ακόμα την οδηγία ε, γι' αυτό στην ομοθεσία τους και αυτό λοιπόν είναι στο χέρι τους να διορθωθεί. Τώρα, ε, σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε τα κονδύλια να δαπανώνται με χρηστό τρόπο, αλλά και όχι μόνο αυτό, και αποτελεσματικά. πρέπει να δούμε και τους ε, ρυθμούς απορρόφη, τα ποσοστά απορρόφησης σε ορισμένα κρατημέλη. Σε κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Στην Ουαλία, για παράδειγμα, το 60% των, των ποσών από τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν απορροφηθεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε οι περιφέρειες των κρατών μελών που έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απορρόφησης να το βελτιώσουν αυτό και επίσης να δούμε τα αποτελέσματα μετά από την ε, πάροδο του χρονικού διαστήματος απορρόφησης. Δεν πρέπει να νομίζουμε πως είναι κάτι απλό, πρέπει να το κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή, να επιβραβεύσουμε τις ε, καλές πρακτικές και να διορθώσουμε τα προβλήματα. Όταν έχουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο μπροστά μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ καλή γνώση του τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχιση του προγράμματος. Είναι ζωτική σημασία στο πρόγραμμα αυτό να έχει καλά αποτελέσματα για να επιβιώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόμασιτς, είστε επόμενη και ο Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τη γνωμοδότησή σας. Υπάρχουν μερικά σημεία μάλιστα που με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι εκεί που ενθαρρύνεται, παροτρύνεται την Επιτροπή και την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου να δώσει ιδιαίτερη βάση στην αναθεώρηση των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και να προσέξουν τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, να τους απλουστεύσουν και Επίσης, συμφωνώ με το σημείο που ζητάτε από την Επιτροπή να δώσει διευκρινήσει στο θέμα του φόρου προς τη αξίας και πώς αυτό μπορεί να επιστραφεί από, το, στην περίοδο, από την περίοδο 2014-2020. Στην περίοδο αυτή ήταν λιγό, λιγότερο από το 20% των εθνικών ε, αρχών είχαν θέτει επιδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να επισπεύσουμε την διαδικασία. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2016 είδαμε ότι δεν είχαν μεταφέρει όλα τα κράτη-μέλη στην νομοθεσία του στην οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες και Χρειάζεται λοιπόν να αυξήσουν τις διοικητικές τους ικανότητες για να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εξαντερεσιμότητας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταμάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η γνωμοδότησή σας για την απαλλαγή σχετικά με τον Γενικό Προβλημό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015 μας επιτρέπει να επανέλθουμε σε κάποια θέματα πιο σημαντικά για την αξιοπιστία της ίδιας πολιτικής συνοχής. Αναφέρονται σε διάφορα σημεία το ποσοστό σφάλματος που εκτιμάται στην πολιτική συνοχή έχει περάσει από 5,7% το 2014 σε 5,2% το 2015 και υπογραμμίζει τις βασικές αιτίες των σφαλμάτων. Θεωρούμε ότι και ένα 5,2% του ποσοστού σφάλματος δεν είναι αποδεκτό και τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Κομισιόν θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να ενδυναμώσουν τα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αποφεύγοντας αυτά που βρίσκονται στην βάση των ε, προβλημάτων, δηλαδή την, ε, την, ε, την εξάρτηση των, μηχανισμών, των ελεκτικών μηχανισμών. Ε, η ταξινόμηση και το reporting των ε, παρατυπιών είναι πολύ σημαντικό και υπογραμμίζω την ουσιαστική σημασία της ισορροπίας που πρέπει να διατηρήσουμε ανάμεσα στην απλούστευση και την, ε, ε, τον διοικητικό έλεγχο. Και υπάρχει μια παράδοση όπου εκφράζεται ανησυχία για το ποσοστό ε, καταβολής για τα 1025 μέσα του ΦΕΣ και του ΕΦΣΕ ήταν της τάξης του 50% 2014, στο τέλος του 2014, μία αύξηση μόνο της τάξης του 10% σε σχέση με το 2013. Θα πρέπει να δούμε ποιοι, ε, ποιοι τομείς και, ποιες, και οι χώρες χρησιμοποιούν τα πετυχάνουν τους στόχους τους, διότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε έτσι την οικονομική, κοινωνική και ε, ταφική πολιτική Συμφωνώ επίση με την Πρόεδρο όταν υπογραμμίζει πως όπως ανέφερε και το Λεκτικό Συνέδριο τη σημασία του να επικεντρωθούμε στι ε, επιδόσεις όπου θεωρείται ευέλικτη πρακτική το γεγονό ότι οι διαχειριστικέ αρχέ καθορίζουν δείκτε αποτελέσματων για να ε, μετρήσουν τον επίτευξη των στόχων που έχουν καθορίσει τα ε, επιχειρησιακά προβλήματα. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποδοτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κ. Λόπες Σάντσες. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία το είπατε το όνομά μου με πάρα πολύ ωραία προφορά. Ναι, είναι πολύ σπάνιο αυτό, λέει ε, η πρόεδρο. Θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω το ίδιο με το δικό σας ε, όνομα, ε, κυρία Μιχαήλοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνετε ειδικότερα να συνοψίσετε στη γνωμοδότηση αυτή, που είναι μία διεξοδικότατη μελέτη του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι μία πρόκληση δύσκολη, έχουμε και εμεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις. Ε, είναι μάλιστα και μία έκθεση ενός ε, ε, μιας ολόκληρης και μακράς ε, χρονιάς ε, ελέγχων. Όσον αφορά στην απαλλαγή αυτή καθεαυτή, που είναι και ο πρώτος λόγος για τον οποίο ερχόμαστε εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντική η άποψη της γνωμοδότης της Επιτροπής σας, του ελεγκτικού συνεδρίου και τον τρόπο, για τον τρόπο, ενδιαφερόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρετε τις απόψεις σας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα ήθελα να ε, αναφερθώ ε, στα διάφορα, σημεία της εκθεσής σας. Μερικά είναι πολύ θετικά, μερικά άλλα είναι λιγότερο θετικά και είναι αμοιβαίο το ενδιαφέρον μας και οι ανησυχίε μας για τα σημεία αυτά. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις για τη βελτίωση της γνωμοδότησής σας. Θα αρχίσω με το πρώτο που είναι θετικό, γιατί εδώ λέτε ότι το ποσοστό σφάλματος έπεσε από τα 5,6, 5,7 είχαμε εμείς υπόψη μας, στο 5,2 το 2015 και λέτε ότι αυτό είναι μία απεικόνηση μιας δεδομένης χρονικής στιγμής. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι η ανάλυση της τάσης και η τάση είναι πάρα πολύ θετική. Όλο και περισσότερο μειώνεται το ποσοστό σφάλματος και αυτό είναι βέβαια πολύ σημαντικό όταν φτάνουμε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του 7-13 γιατί τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να δείξουμε ότι ο ποσοστό, το ποσοστό αυτό ε, σφάλματος ε, ε είναι, έχει μειωθεί κατά το ίμιση ήδη το 2013, το 2013 σε σχέση με το 2006 και νομίζω ότι θα ήταν ε, χρήσιμο σε αυτή τη γνωμοδότηση να το τονίσετε ακόμη πιο θετικά αυτό. Ε, όχι απλώς να λέτε ότι σημειώνουμε με ικανοποίηση, με γιατί αυτό είναι ένα πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αυτή η εξέλιξη και αυτή η τάση μείωσης του ποσοστού σφάλματος. Ε, νομίζω ότι αυτό ε, δίνει πολύ ε, καλό μήνυμα εν αναμονή ε, της ολοκλήρωσης που θα γίνει κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα. Ε, Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό σφάλματος παραμένει ψηλό όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτό το ποσοστό σφάλματος υπολογίστηκε πριν γίνουν όλοι οι έλεγχοι από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατά την ολοκλήρωση λοιπόν του έτους ε, μπορεί να μειωθεί κι άλλο το ποσοστό σφάλματος σε ένα επίπεδο που θα μας επιτρέπει να κλείσουμε το πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν είναι μια απεικόνηση μιας δεδομένης χρονικής στιγμής και όχι τα τελικά ποσοστά. Ε, ε, ήδη το συμπέρασμά σας εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερο, θα το εκτιμούσα ακόμη περισσότερο αν το καθιστούσατε και λίγο θετικότερο. Κάποιο, ένα ακόμη θετικό στοιχείο αφορά το δεύτερο σημείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας, ε, γιατί το βασικό ε, στοιχείο διαβεβαίωσης για μας είναι η δουλειά των αρμοδίων αρχών, ε, των εθνικών αρχών, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι υπάρχει μεγάλη αλλαγή της, ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των εθνικών αρχών. Για μας αυτό είναι καταπληκτικά νέα γιατί Ξέρετε ότι έχουμε πολύ περιορισμένου ε, περιορισμένους ελεκτικούς πόρους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό ε, το ενιαίο πρόγραμμα ελέγχου που είναι η βασική μας ε, δήλωση αξιοπιστία για την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ελεγκτικό συνέδριο να λέει ότι και τα κράτη-μέλη κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλύτερα πλέον προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα φτάσουν και εκείνα το επίπεδο να μας, δίνει, ε, να μας δίνεται ε, η αξιοπιστία που χρειάζεται, που χρειαζόμαστε και εμείς για ε, την απαλλαγή σε σχέση με τον προπολογισμό. Επίσης, οι πηγές φάλματος δεν είναι κάτι το καινούριο. Εμείς το ε, δουλεύουμε. Στο παρελθόν όμως ε, το θέμα των δημοσίων προμηθειών ε, είχε πολύ ψηλότερο ποσοστό. Τουλάχιστον τώρα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί. Το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες προμηθείες και τα μέτρα που λάβαμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία αυτή και τη διαδικασία ελέγχου των δημοσίων προμηθειών. Στο παρελθόν 40% των σφαλμάτων προέρχονταν από τις δημόσιες προμήθειες. Τώρα είναι 15%. Είναι πολύ λιγότερο λοιπόν. Αυτό είναι και μία τάση ακόμη που πρέπει να επιβεβαιωθεί. Πάω στο σημείο 8 ε, γιατί θα ήθελα να πω και ορισμένα πράγματα για τα λιγότερο θετικά στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ για το Omnibus και για την ε, τον έπαινο ε, για το αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονικό, κανονισμό. Υπήρξαν πάρα πολλές προσπάθειες ως προς αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύθηκε στις 14 ε, ε, Σεπτεμβρίου. Έγιναν λοιπόν όλα τα απαραίτητα βήματα για να πάμε προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και ε, της ευελιξίας όπου είπατε και εσείς. Τώρα όμως το μπαλάκι είναι στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, οπότε ελπίζουμε ότι και ε, εσείς ε, ως Κοινοβούλιο θα ε, εγκρίνετε την πρόταση αυτή και ότι θα είναι δυνατόν πλέον για το κράτος μέλος, για τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τις νέες δυνατότητες στον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό και στον τομεακό κανονισμό, στον τομέα ε, της νέας ευελιξίας, για τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και ελπίζουμε ότι είναι μια διαδικασία που θα στεφθεί με επιτυχία και εδώ αλλά και στο Συμβούλιο για την έγκριση αυτής της πρότασης και βεβαίως έχουμε λάβει υπόψη πολύ σοβαρά τις ε, συστάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Και τέλος ε, το σημείο 9. Εμείς επικροτούμε όχι μόνο την, την προσέγγιση του ελεγκτικού ε, συνεδρίου, αλλά και τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις ε, του 1420 ε, για να ε, δούμε ποιες ακριβώς είναι η, ποια ακριβώς είναι η απόδοση του προγράμματός μας. Τώρα, λίγο λιγότερο θετικό ως προς τις ανησυχίε που μα δημιουργεί. Είναι πάρα πολύ καλό να το συζητούμε αυτό γιατί υπήρξαν συνεδριάσει τη ομάδα υψηλού επίπεδου όλη τη μέρα σήμερα. Σήμερα το πρωί μάλιστα συμμετείχα σε κάποιε από αυτέ. Όλη τη μέρα συζητούσαμε πώ μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τι ελεγκτικές διαδικασίε στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με το ελεγκτικό άχθος, το συζητήσαμε ανοιχτά με τον εμπειρογνώμονα της ομάδας υψηλού επίπεδου και αυτό θα δρομολογήσει συστάσεις, οποίες θα λάβουμε υπόψη και όπως ε, γνωρίζετε ε, η Επίτροπός μου ήταν εδώ σήμερα το πρωί και μετά πήγε ε, εκεί για να συζητήσει τι θα γίνει μετά το 2020. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η ομάδα υψηλού επίπεδου. Ήδη έχει θεσμοθετηθεί στο Omnibus ότι όταν χρειάζεται μπορούμε να εισαγάγουμε στον κανονισμό τις ε, συστάσεις αυτής της ομάδας υψηλού επίπεδου. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν ε, χρειάζονται ε, νομοθετικές αλλαγές και νομίζω ότι είναι ε, σωστό αυτό το ε, σχόλιο σας, ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει την έννοια του επιστρεφόμενου ΦΠΑ την περίοδο 14 έως 20 δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό που ήθελε ο νομοθέτης, που είναι να υπάρχει επιλεξιμότητα υπό συγκεκριμένου όρους. Ε, παρόλα αυτά θα το αποσαφηνίσουμε στα κράτη-μέλη και στους δικαιούχους. Φτάνουμε τώρα στο πιο αρνητικό ε, στοιχείο που είναι οι καθυστερήσεις για την περίοδο από το 14 έως το 20 και εδώ. Αυτό που μπορώ να σας πω και το εξήγησε και η Επίτροπος μου σήμερα το πρωί, μας απασχολούν πάρα πολύ αυτές οι καθυστερήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όμως, και πάλι, το ελεγκτικό συνέδριο μόνο μία απεικόνηση έκανε τη δεδομένη χρονική στιγμή στα τέλη του 2015 για το 20%. Εσείς το λέτε όλοι 20%, το οποίο είναι ε, σοβαρό. Όμως είμαστε σε καλύτερη θέση, έχει παρέθει ε, ο χρόνος, έχουμε φτάσει το 2016, ε, πάνω από το ίμιση του προγράμματος έχει ήδη καθοριστεί. Αλλά υπάρχουν ακόμη καθυστερήσει. Ε, απέχουμε πάρα πολύ από το, την ικανοποιητική κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε κάνει αποσαφηνήσεις προς τα κράτη-μέλη για τα σημεία που ε, θεωρούμε ότι μπλοκάρουν ε, τον προγραμματισμό. Ε, δεν ολοκληρώσαμε τη διαδικασία όπως λέγαμε το 2015 αλλά το δουλεύουμε, το επεξεργαζόμαστε είναι κάτι το οποίο θα αποδώσει σε μεταγενέστερο στάδιο της εφαρμογής γιατί θεωρούμε και χρειάστηκε να, κάνει αυτή, να κάνουμε αυτή την ανάλυση και για το μέλλον γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις πάντως η πρώτη μας εντύπωση είναι ότι αυτό θα εξασφαλίσει και καλύτερη ποιότητα στο μέλλον γιατί τα κράτη-μέλη ε, παίρνουν το χρόνο τους για να προετοιμάσουν τα συστήματά τους, να έχουν στεναρά συστήματα με ισχυρές ε, αρμόδιες αρχές για να μπορούν να εκπληρώσουν τις αιρεσιμότητες που ξέρουμε ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον και να έχουν και ένα σύστημα που συλλέγει όλα τα δεδομένα περί απόδοσης που θα χρειαστούμε για να αξιολογήσουμε την ε, ε, απόδοση επί του προγράμματος. Αυτό είναι μια αλλαγή και τα κράτη-μέλη χρειάζονται χρόνο να το κάνουν. Θα θέλαμε λοιπόν να είστε λίγο πιο θετικοί. Χρειαζόμαστε ε, ε, το στοιχείο αυτό μπορεί να μην γίνεται στο βαθμό και στην ταχύτητα που θα θέλαμε αλλά γίνεται για να υπάρχει καλύτερη ποιότητα μετά κατά το στάδιο της εφαρμογής. Επίσης θα ήθελα ε, λίγη αισιοδοξία να ε, εισαγάγω ότι υπάρχει ε, και ένα θέμα επιλογής. Ε, η, η, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το κράτος μέλος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί κάπως η διαδικασία, αλλά μετά θα πάει πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι οι δικαιούχοι σταματούν την εφαρμογή. Υπάρχει μια επιλογή έργων ε, και προγραμμάτων ε, και οι πληροφορίες που έχουμε είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις προηγούμενες προγραμματικής περίοδου, αλλά πράγματι καθυστερεί η διαδικασία. Και ξέρουμε ποια κράτη-μέλη ε, χρειάζονται βοήθεια. Έχουμε στοχεύσει την υποστήριξή μας προς τα κράτη-μέλη αυτή για να βγουν από το αδιέξοδο και να ξεκινήσει η διαδικασία. Μία ακόμη ανησυχία υπάρχει που αφορά ε, συγκεκριμένα οικονομικά μέσα και το είπατε και εσείς αναφέρεστε μάλιστα και στην έκθεση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου για το 57% στο τέλος του 2015 ε, είναι γεγονός ένα χρόνο μετά έχουμε κάποια ε, στοιχεία πλέον, ένα χρόνο μετά, 57% για το τέλος του 2015. Εσείς λέτε ότι υπάρχει μια αύξηση 10% από το 2014. Τώρα έχουμε περίπου αύξηση 20% από το 2014, ε, τέλος του 2014 μέχρι το τέλος του 2015. Και ε, σύμφωνα με διευκρινήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, μέχρι το Μάρτιο του 2017 μπορεί να προσαρμόσει αυτό το το ποσοστό, οπότε ελπίζουμε ότι από το 57% θα πάμε πιο κοντά στο 100%. Ε, Δεν μπορούμε τώρα λοιπόν να συνεπεράνουμε ότι υπάρχει ένα συνολικό κίνδυνος γιατί το ποσοστό έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Και για να ολοκληρώσω από τη Σουμίου 7 θα ήθελα να σα ε, απευθύνω και ένα αίτημα για την έκθεση γιατί εσείς ε, σημειώνετε τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου για την παράταση της περίοδου ε, επιλεξιμότητας. Ξέρετε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται τη σύσταση αυτή γιατί εμείς είχαμε νομικές διατάξεις ε, ε, που δεν μας έδιναν τη δυνατότητα εκταμίευσης ε, μέχρι το 2017. Συνεπώς, ήδη κατά την ετήσια έκθεση του συνεδρίου το 2014 αναφερόταν αυτό, ούτε το Συμβούλιο ούτε το Κοινοβούλιο είχαν υποστηρίξει τη σύσταση αυτή κατά τη διαδικασία της απαλλαγής. Οπότε, θα περίμενα εμείς έχουμε διατηρήσει την άποψή μας ότι είναι νομικό το ζήτημα. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα δεχθεί τη σύσταση αυτή γιατί δεν είναι νομική βάση. Νομίζω ότι θα αρκεστώ σε αυτά και ευχαριστώ να ακούσω ερωτήσεις. Thank you, thank you very I, I... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη πως το σχέδιο έκθεσης είναι αισιόδοξο, αλλά όχι τόσο όσο είστε εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως όμως το επόμενο έτος, όταν κάποιος άλλος συνάδελφος ε, αναλάβει την απαλλαγή του 2016, να ε, σημειώσει όλη αυτή την πρόοδο την οποία ε, αναφέρατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Θα τις συμπεριλάβω όλες, θα τις εξετάσω με προσοχή. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μόνο ότι η καταληκτική ημερομηνία για τροπολογίες είναι η 12η Δεκεμβρίου το μεσημέρι στις 12. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Πολύ κρύο κάνει σήμερα στην αίθουσα και θα γράψω δύο επιστολές στα γραφεία του Κοινοβουλίου ότι κάνει κρύο και ότι δεν έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Συμφωνείτε, θα με στηρίξετε. Όχι. Καλά τότε. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης από τον εισηγητή κύριο Μαρτζή για την διαχείριση των αλλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Επιτροπή Αλληλείας ε, συντάσσει μία έκθεση δύο πρωτοβουλίας και η δική μας Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει και όρισε εισηγητή τον κύριο Γινούσο Μαρτζή, ο οποίος μας ε, παρουσίασε μία πρώτη ε, εικόνα νωρίτερα αυτό το μήνα. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή το Φεβρουάριο του 2017 και στην Επιτροπή Αλία το Μάρτιο. Να προτείνω λοιπόν καταληκτική ημερομηνία για τροπολογίες για τη γνωμοδότηση 12 το μεσημέρι Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου. Κύριο Μαζί, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως τα θερμά ύδατα των εξόχους κέντρων περιοχών θα μας θερμάνουν την ατμόσφαιρα. Εδώ και 15 μέρες είχαμε μια συζήτηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πλούσια στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Δεν θα επανέλθω σε όλα όσα υπόθηκαν τότε και ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους για τις ε, συνεισφορές τους. Έχετε στα χέρια σας την πρόταση που έχουμε καταθέσει. Υπενθυμίζω την άψογη συνεργασία με την Επιτροπή Αλίας και τον εισηγητή ε, Ρίκ Ρολίστ που στο πλαίσιο της ε, κατάρτισης της έκθεσης αυτής έκανε μια διαβούλευση ευρύτατη των εμπλεκομένων των τομέα της Αλίας, στις, ιδιαίτερα στις εξόχους από τις περιοχές και έτσι ακούσαμε το σύνολο των εμπλεκομένων σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό και τους επαγγελματίες του κλάδου. Στην πρόταση λοιπόν που σας έχει υποβληθεί βασιστήκαμε στα θέματα που αφορούν στην Επιτροπή μας. Δηλαδή, και αυτό το θεώρησα σημαντικό, να στείλω ένα ισχυρό μήνυμα προς ε, τους εθνικούς ε, εμπλεκομένους αλλά και τις τοπικές αρχές ε, προκειμένου να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τον αλληλευτικό τομέα στα επιχειρησιακά προγράμματα διότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα χρησιμοποίησης με καλύτερο τρόπο τα διαφορετικά προγράμματα, προ, προγράμματα για να αναπτύξουν τον αλληλευτικό τομέα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που βαραίνουν τον κλάδο, είναι θεμητά, αλλά ήδη υπάρχουν κάποια εργαλεία που υφίστανται και θα πρέπει οι περιφερειακές αρχές ιδιαίτερα να τα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά και να δείξουν πως η αλία στις περιοχές τους είναι ένας από τους πυλώνες της τοπικής ανάπτυξης. Η έκθεση επίσης υπογραμμίζει και το έχουμε συζητήσει εδώ και 15 μέρες το δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης της αλληλείας σε αυτές τις περιοχές που υπενθυμίζουμε ότι εκπροσωπούν 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή και διαπιστώνουμε όλους τους ε, ισχύοντες κανονισμούς γίνεται αναφορά στους ε, κανονισμούς, στους ρυθμίσεις που είχαν ε, σκεφτεί αρχικά για τον Βόρειο Ατλαντικό, για το Βόρειο Μισφαίριο, για την Μεσόγειο, που καταδεικνύονται ακατάλληλες για περιοχές όπως της Καραϊβικής ή του Ινδικού ωκεανού. Και εδώ επανερχόμεθα στην συζήτηση που αφορά την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 349 προκειμένου να υπάρξουν διευθετήσεις ρυθμιστικές, κανονιστικές θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. Το βασικό ερώτημα για το των ε, αλλίων της περιοχής είναι ότι οι κανονισμοί ε, ε, αξιοδοτούν και επιτρέπουν τον εξοχρονισμό και την ανανέωση των αλληλευτικών στόλων. Υπάρχει μια συζήτηση εδώ και καιρό που διεξάγεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο θέμα και υπάρχει πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ειδικά με το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 349. Πιστεύω πως την πρόταση που σας έχω υποβάλει κάνω μια πρόταση αρκετά ισορροπημένη. Δηλαδή, να αδειοδοτήσουμε τον εξορισμό και την ε, διαδιδότηση των ε, στολίσκων υπό τον όρο το σύνολο των ε, αλλοιωμένων εχθείων να εκφορτώνονται στις περιοχές αυτές. Κάτι το οποίο αφορά στην κοινή πολιτική αλληλεία, διότι ξέρετε ότι οι συλλήψεις αυτών των μικρών παράκτιων και αεροτεχνικών αλλιέων που είναι μηδαμινή σε σχέση με τα αλλιεύματα των ευρωπαϊκών και υπολείπων στόλων εκφορτώνονται σε αυτές τις από ε, απόγειες περιοχές κάτι το οποίο επιτρέπει να δημιουργηθεί μια πραγματική τοπική αγορά, κάτι το οποίο αναπτύσσει την ε, οικονομία και έτσι να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτό ε, το, την, ε, την τρέλα θα έλεγα, αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθημερινά με κάτι και αυτών των νησιών. Αυτή είναι η πρόταση της πρότασης. Επίσης αναφέρουμε το θέμα της συνέπειας και συνοχής των ε, συμφωνιών αυτών Αφήσαμε κατά μέρο πολλά ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά μεν, αλλά πρόκειται να τα εξετάσει η Επιτροπή Αλίας και ελπίζω να λάβω πλευρά συναδέλφων συνεισφορές ε, σημαντικές για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην έκθεση του συναδέλφου Μέντε και Κοπής. Ευχαριστώ σκιώδης τώρα κύριε Γιουλό ονόματος του σκιώδους. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Μάρζη για την παρουσίαση αυτή. Θα μιλήσω στο όνομα του σκιώδου συγγητέα κύριου Πόγκα που βρίσκεται στη Νέα Καλυφωνία που λυπάται διότι δεν είναι παρόν σήμερα. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Πόγκα θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Μάρζη για την έκθεσή του και την ποιότητα αυτής. Ε, στηρίζει φυσικά τα όσα είπατε και τα όσα υποστηρίζετε στην εκθέση σας, αλλά και ειδικά στην αναγκαιότητα εξυγχρονισμού και ανανέωσης ε, των στολίσκων των περιφερειακών περιοχών. Ο κύριος Πόγκα μου είπε ότι θα κάνει κάποιες διευκρινήσεις ε, σε τέσσερα σημεία καταρχήν για να τονίσει τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της ε, αηφόρου αλίας και ε, της, ε, ασφάλειας διατροφής να υπενθυμίσει την σκοπιμότητα για να υπάρξει μια ρύθμιση του, για το αλίας με τις εξόχους, για τις εξόχους από τις περιοχές Τρίτον, για να ληφθούν καλύτερα υπόψη αυτό, τα συμφέροντα των περιφών όταν οι συμφωνίες αλίες μπορούν να συνεχθούν με τρίτα κράτη και τέλος ε, να εκφράσει την επιθυμία την καταπολέμηση της ε, λαθροαλίας, της λαθρέας αλίας και της ε, μη ελεγχόμενης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μάσκο για το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως το έπραξε και ο προλαλής σας, να θα ήθελα να χαιρετήσω την εξαιρετική εργασία του συναδέλφου Σομαρζή. Νομίζω πως η μετακίνηση μιας αντιπροσωπείας τον Δεκέμβριο του 2015 η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αλίας αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Σομάρζη κατέδειξε την ε, αναγκαιότητα να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στον τομέα της Αλίας. Το διακύβευμα με διπλό. Να αρθούν τα εμπόδια για να επιτρέψουμε σε αυτόν τον τομέα να εκμεταλλευτεί το δυναμικό του και να ε, βελτιστοποιήσει τα μέσα που παρέχει ε, προπολογισμό της Ένωσης. Αυτό το κείμενο λοιπόν του εισηγητή μας αποτελεί μια εξαιρετική βάση για τις εργασίες. Επίσης ε, μιλάει για τα πλέον εκτήματα τα οποία παρουσιάζει η ανάπτυξη του τομέα της αλίας ειδικά σε ό,τι φορά την ε, ζώνη Z2 αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν καταδεικνύουν ότι η πραγματικότητα της αλίας στις περιοχές διαφέρουν από αυτές που γνωρίζουμε στην Ήπειρο. Αυτή η σημαντική διαφορά αιτιολογεί την ανάγκη ρύθμισης των, των συστημάτων στην αλία, την τόπια αλία. Φυσικά έχουν επιτευχθεί κάποιοι πρόοδοι κατά τη διάρκεια των διαπραγμάτευσης της σημερινής κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Αλλά Διαπιστώνουμε σήμερα παλά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν ο τομέα αυτό των δραστηριοτήτων δεν παρέχει ε, ε, όλες τις δυνατότητες των κλάδων. Συμμερίζομαι την άποψη ότι τόσο οι ε, τοπικές αρχές όσο και τα κρατημένη θα πρέπει να δεσμευτούν αποφασιστικά και στην στήριξη αυτού του τομέα δραστηριότητα. Η ανάπτυξη τη αλληλεία τη περιοχές μας απαιτεί να δημιουργηθούν τομεί ισχυροί και ε, χρηματοδότηση επενδύσει σε ποιοτικά, ποιοτικές επενδύσεις. Τώρα το θέμα των ε, αλληλευτικών ε, στολίσκων είναι ουσιαστικό ζήτημα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν αναπτυξιακό τομέα η κατάσταση των αλληλευτικών σκαφών ε, είναι πραγματικά θλιβερή. Πολλοί από τους νέους μας καταλήγουν αυτήν την δραστηριότητα διότι οι συνθήκες ασφάλειας δεν είναι διόλου ικανοποιητικέ και ο στόλο δεν παρέχει ασφάλεια. Το αναφέρθηκε το άρθρο 349 της ε, συνθήκες της Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μας δίνει την απαραίτητη νομική βάση που θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε το νομοθετικό πλαίσιο ε, την πραγματικότητα της αλίας ε, στις περιοχές αυτές. Ε, πέραν από την ανακαίνιση των σκαφών θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε φιλόδοξοι και να βρούμε ειδικά μέτρα και εργαλεία που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αλία. Σύμφωνα με τα όσα γίνονται με το γεωργικό ποζέ στην Γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσει η Αλία να βασίζεται σε ένα εργαλείο που θα είναι απόλυτα αφιερωμένο σε αυτήν. Θα ήθελα φυσικά να μπορέσω να καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγητή για την ε, καλή δουλειά του και θα ήθελα να τοποθετηθώ και εγώ και να διευρύνω λίγο το φάσμα των συζητήσεων. Η ομάδα ECR κατανοεί το πρόβλημα των εξόχως απόκεντρων περιοχών, ή την έλλειψη επενδύσεων που οδήγησε σε αυτά τα προβλήματα. Αυτές τις διπλές ποινές, όπως τις ονόμαζαν, οι οποίες προήλθαν από έλλειψη στη χρηματοδότηση της δεκαετίας του 70 και του 80, αλλά και προβλήματα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής στη δεκαετία του 90 και έπειτα. Όμω, η ομάδα ECR έχει κάποιες ενστάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για την λύση που έχει προταθεί, δηλαδή τη χρήση του άρθρου 349 για τις εξόχως απόκεντρε περιοχές. Και να είμαι σαφή. Ε, δεν είμαστε αντίθετοι στους στόχου για συγκεκριμένες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρούμε ότι το άρθρο 349 είναι άδικο διότι καλύπτει εννέα ξεχωριστού τομεί Και ο Γιουνούς και ο συνάδελφος από του Σοσιαλδημοκράτε αναφέρθηκαν εξίσου στην ανάγκη να υπάρχουν εννέα ε, διαφορετικές ε, περιφέρειες. Όμως ε, δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτές. Μπορούμε να δούμε και άλλες περιφέρειες οι οποίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αυτό, από τη χρήση του άρθρου 349, ορισμός του οποίου είναι πολύ περιοριστικός. Γι' αυτό λοιπόν υποπτεύομαι ότι ο ορισμός του άρθρου 349 ίσως είναι προβληματικός για την ομάδα μας. Θα θέλαμε επίσης να ε, σταθούμε στην ευελιξία που προβλέπει το Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Θεωρούμε ότι αυτές οι ε, περιοχές ήδη απολαμβάνουν μεγάλα ποσοστά ενισχύσεων και ε, παρεκκλήσεων οι οποίες ε, οδηγούν σε ακόμα περισσότερα ωφέλη και ε, και μεταχείριση. Και αυτό λοιπόν θα θέλαμε να αναλογιστούμε λίγο το τι συμβαίνει και να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης. Πιστεύουμε ότι ο λόγος που αυτές οι εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο αυτήν την ευελιξία που τους παρέχει το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας είναι οι τιμές των προϊόντων αλληλείαν ε, που οδήγησαν στο να πληγεί πολύ σημαντικά ο τομέας αυτός. Και θα ήθελα να πω παρότι λείπει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι δεν έχει δημοσιεύσει ε, κάποια σχετική μελέτη για τον κανονισμό του 2014, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές οι περιοχές να εξυγχρονίσουν τους αλληλευτικούς τους στόλους. Και χωρίς ε, αυτή την ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε το δικό μας έργο. τώρα, να πω κάτι που το λέμε πολλές φορές στην Επιτροπή, αλλά δεν πάβει να παραμένει σημαντικό. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με αυτές τις κοινότητες των οξόγων σαπόκεντρων περιοχών, έτσι ώστε αυτές να, να δυσφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Να αποτελέσουν μέρος της λύσης, να ενημερώνονται οι πολίτες, να γνωρίζουν για το, τι, για το ποιες δυνατότητες έχουν και να έχουμε καλή συνεργασία με τους τοπικού φορείς. Τέλος, όπως είπα και πριν, Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες από την ομάδα μας σχετικά με την εφαρμογή του νέου ε, προγράμματος PCI, το οποίο θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία χωρίς ε, ορατό όφελος, χωρίς να προσθέσει περαιτέρω ευελιξία, χωρίς να αυξάνει την ε, πιθανή βοήθεια χωρίς να προβλέπει κάποια αντικατάσταση των, των μηχανών του αλληλευτικού στόλου. Γι' αυτό νομίζω πως όταν, αφού είδαμε την πολιτική για την Αρκτική βλέπουμε αυτό. Ελπίζω ε, να ε, έχουμε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάτα. Αυτό που υπογραμμίζει ο συνάδελφος ε, ο Μαρζέ είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τον λόγο. Υπάρχει ο Ινδικός ωκεανό, υπάρχουν ε, κάποιοι λεκάνες ε, και η γεωστρατηγική του θέση συμβάλλει στην ε, παγκόσμια διάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν αληθικοί πόροι εξαιρετικά, εξαιρετικοί και εκεί το 80% της διεθνούς ε, βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή, διότι έχει υπάρξει και εισηγητή για άλλο θέμα για το πρόβλημα αυτών των περιοχών. Συμφωνούμε όλοι για τη χρήση του 349 της συνθήκε για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση την οποία μπορούμε να βασιστούμε. Όπως ε, υπογράμμισε στον έγγραφο εργασία ο εισηγητής της Επιτροπής Αλληλείας, τη γνωμοδότηση του συναδέλφου, με την εξαίρεση ορισμένων μεγάλων αλλιευτικών σκαφών με βάση τις, τα Κανάρια νησιά, η αλλίες αυτές τις ε, περιφέρειες, τις ε, άκρως απομακρυσμένες, ε, είναι πολύ... δεν μπορούν να συναγωνιστούν φυσικά. Αυτά τα, τώρα τα προγράμματα live θα πρέπει να λάβουν απόψη αυτήν την ιδιαιτερότητα. Τώρα, δεν έγιναν απαραίτητε αλλαγέ στη ε, δεκαετία του 70-80 και έχει, υπάρχει γύρανση των σκαφών. Ε, περισσότερες φορέ ε, τα ηλεκτρική στόλη είναι αδρανείς και κοντεύουν να, διαλυθούν και αποτέλεσμα είναι η απουσία της ασφάλειας για τους εργαζόμενους αυτά τα σκάφη. Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές διότι οι από κλειμένε περιοχές ήδη πληγήσεις από υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλές ε, επενδύσεις κινδυνεύουν να ε, επηρεάσουν την ελκυστικότητα ε, των περιοχών αλλά και την παρουσία των αλλιέων για θέμα της αλλίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Uh, now... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κάποιος άλλος το λόγο. Εφόσον όχι, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΑ, κύριο Αρμάντο Αστουρτήλ, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα Ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ που δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω κάπως την έκθεση. Γενικά Πιστεύω ότι είναι μια έκθεση αντικειμενική αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν ε, συμπεριλαμβάνει όπως ε, το ζήτημα για την συζήτηση περί επιδομάτων της, ε, στην Αλία, ειδικά τα επιδόματα και επιχορηγήσεις στα αλληλευτικούς τόλους είναι, είναι δραστηριότητε που έχει λάβει ο ΣΑ, ο ΠΟΕ και η Κομισιόν κατανοεί τις δυσκολίες αυτών των εξόχους αποκέντρων περιοχών, τι γνώριζε εδώ και καιρό, γι' αυτό και είχε ζητήσει σε προηγούμενη μεταρρύθμιση μια καλύτερη μεταχείριση. Σε αυτή την ε, μεταρρύθμιση, νέο κανονισμό του Ταμείου για την Αλία εξετάζει και, ε, και λαμβάνει υπόψη τον προβληματισμό για αυτέ τι περιφέρειε. Βρισκόμαστε σε μια διεθνή κατάσταση όπου το να ε, ανοίξουν με τι ε, βάνες για κάποιε επιχορηγήσει θα πρέπει να, μας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η Κομισιόν δεν αντιτίθεται στα επιχορηγήσεις στην Αλία, αλλά το λαμβάνει υπόψη της στο διεθνές ε, διεθνή Συγγερία. Είναι πάμε επανειλημμένα και στον κύριο Ρόμπουστ που θα είναι εισηγητής ε, στην Επιτροπή Αλίας ότι είμαστε διατεθειμένοι να μελετήσουμε το ζήτημα με τρόπο αντικειμενικό χωρίς ε, προκαταλήψεις και όσο πιο συνεργάσιμη γίνεται για να βοηθήσουμε τον εισηγητή να να συντάξει μια έκθεση η οποία θα βοηθήσει τον αλληλευτικό στόλο. Κύριε Κουσαλής, ευχαριστώ. Mm. Thank you. Thank you very much. Mr. Omarjee, would you like to answer? To answer my question. Merci à vous tous pour euh, vos... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα σχόλια, για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να απαντήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε, κατά πρώτο λόγο. Σας καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τους κανόνες, ε, τους εμπορικούς σε διεθνές επίπεδο, αν κατάλαβα καλά. Δεν είναι κανόνες, λέει ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή Τώρα, πού θα οδηγήσουν αυτές τις συζητήσεις και ποιες ε, θα είναι οι απόψεις εκατέρωθεν, ε, αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι υπάρχει, υπάρχει μια συζήτηση. Καταλαβαίνω, λέει ο κύριος Ομερζέ, και είναι δύσκολο να μην κάνω το παραλληλισμό με αυτό που συμβαίνει στη γεωργία και ε, το γεγονός ότι καθίσταται πιο ευάλωτος ο άλλος πυλώνας, ε, η μπανάνα, η ζάχαρη ε, των άκρος περιφερειακών περιοχών, άκρος απόκεντρων περιοχών, βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι απειλούνται με εξαφάνιση ε, τα προϊόντα που παράγει. Αν θέλουμε λοιπόν 25 χρόνια επένδυσης για την αλληλεία να εξαφανιστούν στις ε, περιοχές αυτές, ε, πρέπει να πούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με την απόδοση που δεν είναι η σωστή. Από, από τη δεκαετία του 90 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στην υποστήριξη του αλληλευτικού τομέα στις περιοχές αυτές και το αποτέλεσμα που διαπιστώνουμε και νομίζω ότι συμφωνείτε είναι μία διαπίστωση μεγάλης ευαισθησίας στο πλαίσιο του τομέα αυτού. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας ε, και αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν ε, να ε, ε, γίνει η διαχείριση των αλλιευτικών σκόρων όπως πρέπει στην ε, από απόκεντρες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς, ε, η... αν, θυμάμαι, είχε πει και ο πρόεδρος Ζούγκερ ό. Ε, όσον αφορά στις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, θα κάνουμε μία τελευταίας στιγμής, έναν τελευταία στιγμής προγραμματισμό για τις περιοχές αυτές, γιατί οι χώρες, οι περιοχές αυτές δεν μπορούν λόγω της οικονομικής τους κατάστασης να περιμένουν 10 ακόμη χρόνια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ε, τις πλήττουν και ελπίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ θα ακούσει τις προτάσεις ε, ε, του συναδέλφου Ροντιούς και των ε, υπολείπων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είναι γεγονός ότι και το ΕΛΚ το λέει αυτό, ότι πρέπει οπωσδήποτε, ε, κάποτε υπήρχε το ποζεΐ της αλίας, ε, ένας ε, κανονισμός βάσης, σαν να υπήρχε ένα, σαν το ποζεή της γεωργίας. Είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και την αλία αυτών, που καταργήθηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής και εμείς ενσωματωθήκαμε στο ε, ταμείο ε, για την αλληλεία. Ε, για να μπορέσουμε Τώρα να μπορέσει να αναβιώσει το ποζέι, θα δω και τις σχετικές τροπολογίες. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ε, το περιεχόμενο, γιατί είναι γεγονός ότι έχουν γίνει αλλαγές, όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση ακόμη από τον τελικό στόχο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τα προσκόμματα τα που υπάρχουν ε, στην ανάπτυξη του αλλιευτικού τομέα στο, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Πολλά ε, ερωτήματα δεν ετέθησαν, γιατί προφανώς έχουμε έναν αριθμό χαρακτήρων Ω περιορισμό στη γνωμοδέτηση. Γι' αυτό ακριβώ οι τροπολογίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα εμπλουτίσουν αυτήν την έκθεση. Ξέρω την άποψη του ECR για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ε, πιστεύω όμως ότι υπάρχει μία αντίφαση. Αν πιστεύετε ότι ε, Ε, η δυνατότητα που δίνεται από το άρθρο 340 ε, για τις ε, παρεκκλήσεις που αφορούν τις εξώκωσες από έκεντρες περιοχές, ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστείτε το στόχο σας αυτό που είναι η επέκταση του 349 είναι ακριβώς αυτή. Πρέπει να υποστηρίξετε το 349, όχι να το πολεμάτε, γιατί δεν θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε την ε, διεύρυνση που θέλετε. Το άρθρο 349 στόχο έχει τις περιοχές που είναι εξορισμού άκρος απόκεντρες. Είναι πάρα πολύ μακριά από την Ήπειρο και λόγω αυτού αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες για να μπορέσουν ε, ε, να συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά, ε, έχουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωση, τη μεγάλη απόστοση, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν ιδιαίτερη μεταχείριση. Όμως ε, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αγνοεί στους κανονισμούς της ε, τις ιδιαιτερότητες των υπολείπων ευρωπαϊκών περιοχών. Υπάρχουν στρατηγικές οι οποίες εφαρμόζονται για τις ορεινές περιοχές, για τις νησιωτικές περιοχές, για τις άρεοκατοικημένες περιοχές. Όμως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές Ξέρετε, ας πούμε, η Ρεουνιόν είναι σε 10, στα 10.000 χιλιόμετρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προβλήματα ε, τα οποία είναι μόνιμα λόγω, ε, με μειονεκτήματα που είναι μόνιμα λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ε, είναι κάτι το το να λέμε δηλαδή ότι θα πρέπει να πληγούν αυτές οι περιοχές λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της απόστασή τους από ε, οποιοδήποτε από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ε, αναμένω λοιπόν την υποστήριξή σας. Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα σας θα έχει προτάσεις οι οποίες, τις οποίες θα μπορέσω να αποδεχθώ και το ίδιο ισχύει και για τον συνάδελφο ε, Λουί Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες μεσημέρι Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα συντάξει μια έκθεση βίας πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή της Επενδύσεων και τον έλεγχο των ε, δραστηριοτήτων της για το 2015. έχει αυξηθεί η δράση της τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και αναμένεται περαιτέρω αύξηση. Ο εισηγητής κ. Γιάκοφτσι σήμερα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Προτείνω την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι να είναι καταληκτική ημερομηνία για υποβολή τροπολογιών και θα δώσω το λόγο αμέσω στον κύριο Γιάκοφτσιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχής να σα ε, ζητήσω να κάνετε ό,τι μπορείτε να παρατείνουμε λίγο την καταληκτική ημερομηνία τροπολογιών για τις 20 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα που συναντήσαμε και θα χρειαστούμε μια παράταση. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα, ε, διότι δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες εργασίας μας σε αυτή την αίθουσα. Εντάξει, εγώ βέβαια μπορώ να αντέξω το κρύο γιατί έχω κάποιο ειδικό βάρος, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Συντομότερος από ό,τι υπολόγισα. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να πω πως χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να συντάξω αυτή τη γνωμοδότηση και ευχαρίστως να λάβω υπόψη όλες τις ιδέες και τις προτάσεις σας για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τώρα και στο μέλλον. Να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι τώρα έχει επενδύσει 77,5 δισεκατομμύρια σε υποδομές, στο περιβάλλον, σε καινοτομία, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει επενδύσει μόλις 7,5 δισεκατομμύρια. Ε, και αυτό πρέπει να δημιουργήσει όμως κάποια συνέργεια όταν θα αρχίσουμε να εξετάζουμε το ποιος έχει ανάγκη τα κονδύλια. Τώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανομή των ε, κονδυλίων στους ε, κύριους ε, δικαιούχους ήταν, μάλλον πήγε στους μεγάλους, στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Γερμανία. Και τα νέα κρατημέλη έλαβαν λιγότερο από το 20% των κονδυλίων. Αυτό δείχνει ότι και τα κράτη-μέλη χρειάζονται τεχνική βοήθεια και περισσότερες ευκαιρίες. Πρέπει και τα ίδια να γίνουν πιο δημιουργικά για να μπορέσουν να ζητήσουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γι' αυτό βλέπω εδώ πως υπάρχει ανάγκη για συνέργειες ανάμεσα στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την ΕΤΕΠ ή και μετά διαρθρωτικά ταμεία, όπως στο παρελθόν. Διότι θεωρώ πως αυτή η συνέργεια θα οδηγήσει στην αύξηση της ποιότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων οφείλει να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα. Να τονίσω επίσης και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια Βουλγαρία, Ιταλία, Φιλανδία, Μάλτα, Ρουμανία, Ισπανία και Κροατία είναι χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν αυτά τα ποσά και είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούν να συνεισφέρουν πολύ θετικά στην ανάκαμψη της οικονομίας αυτών των χωρών ή στην ε, βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω και από τους συναδέλφους της ΕΤΕΠ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να μας στηρίζουν, να στηρίζουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, διότι και εκείνες συμμετέχουν στην ανάπτυξη ορισμένων περιοχών. Εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, γνωρίζουμε το τι συμβαίνει, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να στηρίζει κανείς τις τοπικές αρχές. Και κάτι άλλο. Να πω ότι θα ήταν καλό, πέρα από τα μέσα διασυνοριακής συνεργασίας, να δημιουργούσαμε μέσα για μακροπεριφερειακή συνεργασία. Υπάρχουν ήδη κάποια προγράμματα για το δούναβη, για τη Σάλπη, τη Βαλτική, τη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει όμως κάποιο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο θα μπορούσε να καλύψει 5-6 χώρες ε, μαζί στα πλαίσια μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Και αν δεν δώσουμε προσοχή σε αυτό θα δαπανίσουμε πολύ κόπο και χρόνο για όχι καλά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο χρηματοδότησης. Δεν θα μιλήσω άλλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ε, να πω πως είμαι σίγουρος για μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στο ο κύριος Βάλκαρσελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια για να συγχαρώ τον κύριο Γιάκοβιτς για την εργασία του. Φυσικά το ζήτημα που τον απασχόλησε, μάλλον που, ε, αφορά στην ε, ΕΤΕΠ, ε, γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Αυτές οι δραστηριότητες, αυτές οι πράξεις είχαν σαν αποτέλεσμα να βελτιώσουν την διοικητική ικανότητα αλλά και τη δημιουργία συνέργειας ε, ανάμεσα στα ταμεία όπως ανέφερε και ο εισηγητής. Επίσης θεωρώ ε, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθήσουμε τους σύναγκες στην πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι με αυτήν την όθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βλέπουμε πως η οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί και οι επιπτώσεις οι άμεσες ε, που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και φέρουμε και πολιτικές ευθύνες ε, είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες προκειμένου να συμβάλλω αλλά και να προσπαθήσω να εμπλουτίσω το λέω με κάθε μετριοπάθεια το κείμενο το οποίο αυτό καθε αυτό είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λούρα έχει το λόγο, επόμενος και ο δυσήγητης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Θα χαρώ να συνεργαστούμε. Εντάξει, μπορεί να φταίνε τα 25 λεπτά που περίμενα στην παγωνιά, αλλά εγώ δεν νιώθω κρύο εδώ, δεν κρυώνω. Αλλά εντάξει, θα είμαι κι εγώ σύντομο. Η ομάδα ECR στηρίζει σε γενικές γραμμέ την ε, στήριξη της ΕΤΕΠ, ιδιαίτερα αφόσον μετά την ε, οικονομική κρίση του 2008 δεν ε, χρειαζόμαστε περισσότερους ε, πόρους. Χρειάζεται να δώσουμε μία όθηση στην ανάπτυξη. Όμως η ομάδα ECR δυστυχώς είδε ότι υπήρξαν προβλήματα, υπήρξε αύξηση των καθυστερήσεων το 2015 και εμείς, να είστε σίγουροι, θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις για την έκθεση του 2016. Τώρα, πέραν αυτού, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να βρούμε συνέργειες ανάμεσα στη, στην ΕΤΕΠ και στο ΕΦΣΥ. Η ομάδα μας, λοιπόν, θα συνεχίσει να ζητά από την ΕΤΕΠ να συνεργάζεται όποτε μπορεί με τις αρμόδιες αρχές και να οδηγηθεί στην, ε, στη δημιουργία συνεργειών. Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε αυτά να συνδυαστούν με τις πρωτοβουλίες που αναφέρατε δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένους ε, ορισμένους, ε, ορισμένες συνεργασίες, ιδιαίτερα μάλιστα τώρα σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να διασφαλίσει ότι θα χρηματοδοτήσει προτάσεις και έργα που θα έχουν προστιθέμενη αξία και να φροντίσει να μην επιβαρύνει άλλο τους προπολογισμού των ε, κρατών μελών. Ε, επίσης πρέπει να μιλήσουμε και για τη γεωγραφική κατανομή των ενισχύσεων. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία συνεισφέρουν στο πάγιο κεφάλαιο της ε, Τράπεζας Επενδύσεων και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στόχο έχει να στηρίζει οικονομικά ε, αδύναμες οικονομικά περιοχές εκτός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει κάνει με την Ουκρανία για παράδειγμα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πολύ ισχυρό ε, αδιάβλητο χαρτοφυλάκιο ενισχύσεων και η έλεγχη να είναι εξονυχιστική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο, να πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεισφέρει τα μεγαλύτερα ποσά στην ΕΤΕΠ και δεδομένου του αβέβαιου μέλλοντος μετά το Brexit πρέπει να διασφαλίσουμε οι βρετανικές αιτήσει να αξιολογούνται αντικειμενικά. καθώς εμείς θα προσαρμοζόμαστε στη νέα μας πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βόν, θα θέλατε το λόγο, είστε και εσείς και ο Ναι, σας ευχαριστώ. Να πω καταρχάς ότι όλοι στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Πιστεύω όμως ότι η Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να ε, γίνει χρηματοδότης. Ε, τα, περισσότε, τα περισσότερα κονδύλια προέρχονται από επιχορηγήσεις. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να αλλάξουμε το, τα ποσοστά αυτά, να αλλάξουμε τα νούμερα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά προγράμματα που στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Έπειτα πρέπει να διασφαλίσουμε την δημιουργία συνεργειών. Η ΕΤΕΠ έχει κάποιες ε, καλές εμπειρίες από το παρελθόν, έχει χρηματοδοτήσει κάποια καλά προγράμματα, εκπαιδευτικά, ε, προγράμματα σε πανεπιστήμια αλλά έχει συνεργαστεί και με τα διαρθρωτικά ταμεία έτσι ώστε να συγχρηματοδοτήσουν προγράμματα. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα αυτής της συνεργασίας και πρέπει να την ε, ε, ενθαρρύνουμε για να συνεχιστεί στο μέλλον. Τώρα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα είχαν και κάποια προβλήματα. Έλειπε κάποιος σχετικός δημοσιονομικός κανονισμός. Έχουν αρχίσει να γίνονται βελτιώσεις, πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι τα κονδύλια είναι πολύ ψηλά, υπάρχουν ποσά τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί και πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί. Πρέπει να δούμε και τον αριθμό των έργων που χρηματοδοτούνται, τον αριθμό των αιτήσεων, διότι πιστεύω ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε αλλά και πολλά να χάσουμε αν δεν το κάνουμε αυτό πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να τοποθετηθεί ιδιαίτερα για το θέμα αυτό των υπέρογκων ταμείων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταμάτο. Σχετικά με τη γνωμοδότηση για τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ για το 2015 έχουμε κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με την αύξηση του κινδύνου και την μετακίνηση σε προς ειδικά ειδικά χρηματοπιστωτικά μέτρα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να αλλάξουν εδώ κάποιοι μηχανισμοί δημοσιονομικοί που θα οδηγήσουν σε ένα αυτεπίστροφο. Αντί να ε, ε, ωφελήσουμε το κλίμα, τους επενδυτές ε, για... και να τους δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο κλίμα. Υπάρχουν προγράμματα όπως το ΤΑΡ στην Ιταλία έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Πολλές παρεμβάσεις εξάλλου δεν αποκρίνονται στους στόχους της ε, μείωσης ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει και το ζήτημα του μετρό του Μιλάνου που ε, έχει εμπλακεί στο ζήτημα και το οργανωμένο έγκλημα και η έμεση χρηματοδότηση υπέρ των οικονομικών επιχειρήσεων συχνά βασίζονται σε κεροσκοπικά κεφάλαια που δεν ακολουθούν τον στόχο της ενδυνάμωσης της πραγματική οικονομίας. Σε ό,τι αφορά επίσης τη δέσμευση της τέ για το ΕΦΣΥ, διαπιστώνω για μια ακόμα φορά με απογοήτευση την στήριξη ε, χαλιβουριών, ε, Αποθήκευση αερίου όπου το 5% των ε, επενδύσεων του ΕΦΣΙ αφορούν ε, ε, τους ορυκτές, τα ορυκτά καύσιμα. Κάτι ακόμα θα πρέπει να προσέξουμε, όπως η δέσμευση της ΕΤΕΠ υπέρ της, των ανανεώμενων πηγών ενέργειας. Και ενώ, συνεχίζει να, κατασκευάζει τα τεράστιες καταστάσεις ε, αιωλικών, ε, αιωλικής ενέργειας δεν, ε, δεν κάνει συγχρόνως και τα παράλληλες επενδύσεις σε άλλους εξίσου σημαντικούς για την ενέργεια κλάδου Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν δεις άλλους να λάβει τον λόγο, δίνει τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ρίτσο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ τους αξιότιμους ευρωβουλευτές. Ε, ε, όσον αφορά τα ε, υπέρογγα χρήματα πιστοτικά ε, ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επιπλέον σχόλια παντό στον κύριο Βον. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την καταληκτική ημερομηνία για τις προθεσμίες 7 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι και τώρα να σας δώσω το λόγο. Κοιτάξτε, ρώτησα στην αρχή αν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο την ε, ημερομηνία υποβολής μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Ξέρω, ξέρω ότι τεχνικός γίνεται αυτό και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μας αν μπορείτε να το κάνετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εξέφρασαν την υποστήριξή τους για αυτήν την έκθεση. Σε σχέση με το Brexit ε, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι μεγάλος επενδυτής στην ΕΤΕΠ, οπότε συμφωνώ με την προσέγγισή σας. Ε, ίσως θα μπορούσαμε και για το 2015 να συμπεριλάβουμε ε, μία ε, έκθεση. Όσον αφορά τα προγράμματα ενεργειακής υποδομής, είναι σημαντικό να μιλούμε για, πηγές, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να τονιστεί, γιατί είναι μία από τις προτεραιότητες της ΕΤΕΠ. Αυτά από μένα. Αν μπορούσατε μόνο να ε, απαντήσετε το ερώτημά μου σε σχέση με την παράταση της ημερομηνίας ε, κατάθεσης τροπολογιών. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μέχρι τι 7 Δεκεμβρίου θα θέλαμε τις, προθε... Ε, τροπολογίες για να μπορέσουμε να τις μεταφράσουμε πριν τα Χριστούγεννα και να μπορέσουμε, ε, επειδή ακριβώ έχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, ε, καλό θα ήταν ε, για τους ε, σκιώδει εισηγητές. Εντάξει, εντάξει, λέει ο κύριος Γιάκοφτσιτ. Δυστυχώς κλείνει το μικρόφωνο της Προέδρου και δεν ακούμε. Λοιπόν, έχουμε σχεδόν παγώσει μέσα σε αυτή την αίθουσα. Έχουμε κάτι ακόμη να κάνουμε και μετά θα έχουμε αφήσει τα κοκαλάκια μας στην αίθουσα. Κύριε Βανίστελ Ρόι, μήπως μπορείτε να μας παρουσιάσετε το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για την προφορική ερώτηση που συζητήσαμε ε, στην συνεδρίαση των συντονιστών. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, πολύ σύντομα. Ο στόχος αυτού που κάνουμε είναι ε, αυτή η ανησυχία της Επιτροπής μας που έχει εκφραστεί ε, σε άλλα έγγραφα την εκφράζουμε στην Ολομέλεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν βλέπουμε τον προϋπολογισμό για το 2017 υπάρχουν συμπεράσματα του Συμβουλίου, δηλαδή για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός μας ε, είναι 24% χαμηλότερος ε, από ε, τον αρχικά προβλεπόμενο. 7,3 δις λιγότερα και αν δει κανείς ε, το 2009 την τελευταία περίοδο από το 2009 το 2014, συγγνώμη, 2007 με 2014, αν δει, πώς, ε, αν δει κανείς πώς έχουν τα πράγματα τώρα, είναι πολύ σοβαρότερη και βαρύτερη η κατάσταση, είναι πολύ λιγότερη η αποδοτικότητά μας, ε, αποδοτικότητά μας σε σχέση με το παρελθόν. Αν δει κανείς τα αριθμητικά στοιχεία, ε, θα το καταλάβει αυτό. Καλό θα ήταν να το συμπεριλάβουμε αυτό στο κείμενο για να μπορέσουμε να ε, το θέσουμε. Είναι σημαντικό η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να το κάνει τώρα και όχι την επόμενη χρονιά, γιατί ήδη η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα αρχίσει να δουλεύει ε, για τους επόμενους προϋπολογισμούς. Ε, είναι δική μας η πολιτική αυτή. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε έργο ή αλλιώς θα τιμωρηθούμε. Έχουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις λοιπόν ως προς αυτό και έχω ένα κείμενο το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση ε, και να λέει ότι εμείς ε, δεν είμαστε ε, η γαλοπούλα των Χριστουγέννων, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να έχουμε, να, έχουμε την κύρια άποψη βάσει της οποίας θα ληφθούν οι αποφάσεις και εμείς θα πάρουμε την μπάλα πρώτη για να το πω έτσι. Ε, αυτές βέβαια οι προτάσεις μπορούν να βελτιωθούν, να αλλάξουν. Ε, ε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Είναι ένα πρώτο κείμενο αυτό για το ψήφισμα. Ένα ψήφισμα το οποίο θα έχει προέλθει από εμάς. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε ήδη πει ότι θέλουμε να συνεργαστούμε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το έχουμε ξανακάνει αυτό. Ίσως το Φεβρουάριο να κάνουμε μία συζήτηση για το άρθρο 16.3 ε, κάποια στιγμή και να μπορέσουμε να έχουμε μια ε, συγκεκριμένη, να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτά. Ευχαριστώ, όχι εμείς δεν είμαστε η γαλοπούλα των Χριστουγέννων, παρόλα αυτά μπορούμε να είμαστε κατεψυγμένοι γαλοπούλα. Ίσως αυτός ε, είναι ο λόγο αυτού του κρύου στην αίθουσα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή. Κοιτάξτε, τι προτείνω για το χρονοδιάγραμμα για αυτό το θέμα. Σήμερα έγινε η παρουσίαση του σχεδίου ψηφίσματος στις 13 Δεκεμβρίου. Ε, θα διανεμηθούν οι μεταφράσεις σε όλες τις χώρες. 19 Δεκεμβρίου θα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Το Στρασβούρ, στο Στρασβούργο τον Ιανουάριο μπορεί να γίνει μια συνάντηση των σκιωδών για να συζητήσουμε το σχέδιο ψηφίσματος και το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος και μετά μπορούμε να ψηφίσουμε το, ε, το ερώτημα και την ε, πρόταση ψηφίσματος. Αν συμφωνείτε μπορούμε να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό διάφορα. Σας παρακαλώ, μην έχετε διάφορα, κάνει πάρα πολύ κρύο. Να σας υπενθυμίσω τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Ε, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 6 και μισή και 24 Ιανουαρίου όλη την ημέρα. Εδώ Κλείνω τη συνεδρίασή μας, τουλάχιστον το δημόσιο τμήμα της συνεδρίασης και συνεχίζουμε και κλεισμένων των θυρών ε, με τους συντονιστές. Είναι εδώ κανείς που δεν είναι συντονιστής? Μπορούμε να κάνουμε γυμναστική, προτείνει ο κύριος Φανίστελ Ρόι, για να μην κρυώνουμε.